Καλημέρα, συνάδελφοι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Πρέπει να ξεκινήσουμε τι εργασίε μα. Και ακόμα και αν δεν είμαστε πλήρεις, πρέπει να προχωρήσουμε στον αφορά την ημερήσια διάταξη. Και να ακούσαμε και τις παρεμβάσεις και των εμπειρογνωμών που καλέσαμε αλλά να ακολουθήσει και δέουσα συζήτηση επί ενός άκρου ενδιαφέρου ενδιαφέροντος θέματος όπως είναι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το Συμβούλιο Συνεργασίας των χωρών του κόλπου. Αυτή η συνάντησή μας προηγείται των εκθέσεων που ο συνάδελφος αντιπρόεδρος Ντομινίκ Μποντής θα ετοιμάσει μαζί με τον κύριο Μάριο Ντάβιντ που είναι εισηγητή επί του θέματος για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Είναι αρκετά παράδοξο το ότι αυτή η περιφέρεια του κόσμου, η περιοχή του κόσμου, που είναι τόσο σημαντική από πλευρά στρατηγική και λόγω της τοποθεσίας, είναι σε μια κεντρική περιοχή όσον αφορά τα προβλήματα που πλήττουν τη Μέση Ανατολή και τόσα χρόνια αυτή η περιοχή δεν έτυχε της δέωσας προσοχής και πολιτικής ε, αξιολόγησης. Λοιπόν, προστίθεται σε αυτό το πλαίσιο και το εξή, ότι εδώ και 20 χρόνια προσπαθούμε να συνάψουμε με το Συμβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, κάτι που δεν συνέβη ακόμα παρά το ότι είναι η μεγαλύτερη αγορά, η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά όσον αφορά τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος αυτών των χωρών. Όλα αυτά τα θέματα μαζί με το γεγονός ότι έγιναν σημαντικές κοινωνικές αλλαγές και αλλαγές στους πολιτικούς θεσμούς αυτών των χωρών, όλα αυτά αξίζουν την προσοχή μας και την υποστήριξή μας χρειάζεται να ασκηθεί μια πιο φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά αυτή την στατηγική περιοχή. Θα πρέπει να προωθηθούν τα κοινά συμφέροντα περαιτέρω, να δημιουργηθεί χώρο σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και να δημιουργηθούν οικονομικοί δεσμοί πιο στενοί και πιο εντατικοί. Και αυτή είναι επιθυμία και ευχή και για αυτούς τους λόγους συναντώμεθα πάνω σε αυτά τα θέματα με τους εμπειρογνώμονες που έχουμε προσκαλέσει. Οι εμπειρογνώμονες θα μας βοηθήσουν να εξετάσουμε το θέμα. Ο Dr. Christian Koch, ο κύριος Christian Koch, διευθυντής για τις εξωτερικές, εξωτερικές σχέσεις του Κέντρου Ερευνών για την περιοχή του κόλπου και ο κύριος Ζωζιέ Φιλίπ Μπερτότσι που είναι διεθνής σύμβουλος και εμπειρογνώμων όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Συμβουλίου των χωρών της περιοχής για τη συνεργασία με τις χώρες του κόλπου. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Κοκ και τον παρακαλώ αν μπορεί να συγκρατηθεί χρονικά σε ένα δεκάλεπτο αν μπορεί όσον αφορά την παρέμβασή του. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτρέψτε μου καταρχά να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τη δυνατότητα που μου δίδεται να εμφανιστώ εδώ και να αναφερθώ στι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασία των... του Κόλπου. Πάνω από 20 χρόνια πέρασαν από τη στιγμή που εγγράφει η Συμφωνία Συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και του Συμβουλίου Συνεργασία των Χωρών τη ε, περιοχή του Κόλπου τον Ιούνιο του 1988. Αυτή η συμφωνία μα έχει δημιουργήσει το πλαίσιο για την αμοιβαία ε, εποφελών σχέσεων και επιτεύγματα, τα επιτεύγματα της συμφωνίας όμως απέχουν των προσδοκιών. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις δεν αναπτύχθηκαν καθόλου, ότι υπάρχουν ε, διάφορα προβλήματα και εμπόδια που δεν μπορούν να έρθουν ή ότι υπάρχουν προβληματικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια, είδαμε να επανέρχεται το πνεύμα της Συμφωνίας για τη Συνεργασία του 1988 με επιθυμία να ενισχυθούν και να εφαρμοθούν οι θεσμικοί ε, δεσμοί. Και αυτό είναι οραστό στην υιοθέτηση της, ε, του κοινού προγράμματο που υθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο των Χώρων τη Περιοχή, των Υπουργών τη Περιοχή, και είναι ο δικό χάρτη για να αναπτυχθούν οι σχέσει σε 14 συγκεκριμένου τομεί. Και όσον αφορά τι διαπραγματεύσει για τη ζώνη ελευθερών συναλλαγών που έχει επικριθεί, οι συνομιλίε που διεξήχθησαν από το 2003 στο 2008 μπόρεσαν να πετύχουν σημαντική πρόοδο και οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ κοντά στην ολοκλήρωση, διεκπαιρέωση των συμφωνιών και να καταλήξουν να καρποφορεί συμφωνία. Επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ το κοινό πρόγραμμα δράση σε σημαντικό βήμα προ την κατεύθυνση. Όμω πιστεύω επίση ότι το σχέδιο δράση υπολείπεται ε, των στόχων σε δύο σημαντικού τομεί. Πρώτα απ' όλα, καταρχά, παραμένει απλώ ένα προσανατολισμό για το πού ελπίζουμε ότι κατευθύνουν οι σχέσει και δεν παρέχει δεν προβλέπει συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή των διαφόρων τομέων συνεργασίας. Παρά την ανακοίνωση που έγινε για τους διάφορους μηχανισμούς που θα έπρεπε να εφαρμοστούν μέχρι το 2013, κάτι που επιτάσσει συμφωνία, δεν είδα συγκεκριμένα βήματα. Δεύτερον και πιο σημαντικό, οι, πολιτικ... οι πτυχέ πολιτική και ασφαλεία όσον αφορά τι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ενώση με αυτή την περιοχή του κόσμου δεν αναφέρονται καθόλου. Αυτό είναι κρισίμου σημασία, διότι αν κάποιο πιστέψει ότι είναι φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να γίνει σημαντικό πολιτικό φορέα στην στατική περιοχή του κόλπου, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετό για να καθορίσει κανείς τις σχέσεις με τις χώρες ε, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ε, διότι από αυτή την προσέγγιση θα βασίζονται μόνο στην ενέργεια, στην οικονομία και στο εμπόριο. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα θέματα και ερωτήματα, γιατί πρέπει να προσέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα όσα τεκταίνονται στην περιοχή του κόλπου γιατί θα πρέπει η ανάπτυξη σχέσεων με τις χώρες του κόλπου να είναι η βάση μία αναζωογονημένης συνεργασίας και εταιρική σχέσεω και ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι τομεί στου όποιου μπορούν να γίνουν συγκεκριμένα βήματα και να πετύχουν συγκεκριμένα πράγματα. Στο πρώτο ερώτημα, γιατί είναι σημαντικό ο κόλπος για την Ευρώπη. Εάν συνδυάσουμε τις διάφορα χαρακτηριστικά που ε, συναθρίζουν την εξουσία και την ασφάλεια, δεν υπάρχει σημαντικότερο τμήμα του κόσμου σήμερα από την περιοχή του κόλπου. Γεωγραφικά η περιοχή είναι στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολή και Δύση και συνδέει τι τρει υπήρου τη Ασία, τη Αφρική και τη Ευρώπη. Πολιτιστικό, το βασίλειο τη Σαουδική Αραβία είναι η πατρίδα του Ισλάμ, που είναι μια θρησκεία, η θρησκεία του κόσμου αναπτύσσεται των χείρο ρυθμών. Και η συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τι μουσουλμανικέ κοινότητε και την ένταξη και την ολοκλήρωση ε, είναι ένα θέμα στο οποίο δραματίζει ρόλο η περιοχή. Όσον αφορά την ενεργειακή πτυχή, ο, έχει 60% των αποθεμάτων πετρελαίου ο κόλπος και παρέχει το 1 τρίτο της καθημερινής παραγωγής του πετρελαίου. Καμία άλλη περιοχή στον κόσμο θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου για το πετρέλαιο τις επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες περισσότερο από τον κόλπο. Λοιπόν, οι χώρε του κόλπου καταβάλουν σοβαρέ προσπάθειε, ώστε να αναπτύξουν εναλλακτικέ ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Όσον αφορά το ευρύτερο οικονομικό πεδίο, οι χώρε του Συμβουλίου του Κόλπου είναι σημαντικοί φορεί και όσον αφορά την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και την σταθερότητα όσον αφορά τι παγκόσμιε χρηματοστικέ αγορέ. Σαουδική Αραβία είναι η μόνη χώρα τη Μέση Ανατολή που είναι μέλο ε, των G20 και γενικά ε, πιστεύετε ότι οι χώρε του Συμβουλίου Συνεργασία του Κόλπου θα έχουν ένα πλεόνασμα 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων του 2015 με, με το συνδυασμένο ΑΕΠ θα φτάσουν τα 2-3 το 2020 και ε, τα, έχουν ε, αξιόγραφα που είναι πάνω από 1,3 3 εκατομμύρια χώρε του κόλπου και είναι κρίσιμο σημασία σε πολλού τομεί για την υποστήριξη βασικών βιομηχανιών στα κράτη-μέλη μεταξύ άλλων. Επιπλέον, οι χώρε Συμβουλίου του Κόλπου είναι στην πρώτη γραμμή σχετικά αφορά την βοήθεια ε, σε μακρινέ χώρε και έχουν συμβάλει σημαντικά στη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων και κατεπίκουσα βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Πιο σημαντικό για τη συζήτηση είναι ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η περιοχή του κόλπου είναι στο επίκεντρο όσον αφορά τα θέματα τη ειρήνη και τη ασφαλεία. Όχι μόνο για την ίδια την περιοχή, αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο επίση. Οι εντάσει στον κόλπο εξακολουθούν να έχουν συνέπειε σε παγκόσμιο επίπεδο και οδήγησαν στην συμμετοχή ε, και ανάπτυξη ξένων δυνάμεων στην περιοχή μας δείχνουν οι τάσεις ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη διεθνοποίηση στο μέλλον και ανταγωνισμός όσον αφορά τους πόρους της περιοχής, κυρίως από πλευράς χωρών της Ασίας. Δοθισών αυτών των εξελίξεων η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι στο περιθώριο διότι δεν έχει προσέξει μέχρι τώρα την περιοχή του κόλπου Εξίσου σημαντικό είναι να καταλάβει κανεί τι αρνητικέ συνέπειε για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν συμμετέχει περισσότερο και συνεργαστεί με την περιοχή αυτή. Μερικά παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα, η επίλυση του προβλήματο του προγράμματο του πυρηνικού ε, του Ιράν δεν είναι μόνο κάτι που είναι σημαντικό για την ασφάλεια τη περιοχή, αλλά και για το μέλλον τη μη διάδοση των πυρηνικών προ τον κόσμο. Το Συμβούλιο των Χωρών του Κόλπου δεν θέλει να δει άλλη σύραξη στον κόλπο, αλλά ούτε θέλουν να ζήσουν και στη σκιά ενό ε, εξοπλισμένα με πυρηνικά όπλα Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει κίνδυνο ορατό να υπάρξει ε, άλλο κύκλο Ιράκ στην περιοχή ή να αποκτήσουν τι χώρε τη περιοχή πυρηνικών όπλων. Και η εσωτερική ασφάλεια του Ιράκ επίση ε, δεν εξασφαλίζεται και αυξάνονται εντά στην περιοχή. Περιφερειακέ και διεθνεί προσπάθειε είναι ουσιαστικέ ε, πάρα πολύ σημαντικέ για να μην υπάρξει επιδείνωση στον φάτη σταθερότητα του Ιράκ. Η Εμένη πρέπει να είναι ένα ενωμένο κράτος και να αποφευθεί νέο εμφύλιο πόλεμο και ακρεφνή στοιχεία όπω το δίκτυο τη Al-Qaeda που θέλουν να κάνουν τη εμένη βάση των επιχειρήσεών του σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Σαν μεγαλύτερο γείτονα, τίποτα δεν ησυχεί περισσότερο μια χώρα όπω η Σαουδική Αραβία όταν βλέπει την Ιεμένη να είναι μια χώρα αποτυχημένη και άναρχη. Η σύραξη μεταξύ Λιγνών και Αράβων είναι βασικό πρόβλημα στην περιοχή ε, και που επηρεάζει τα συναισθήματα όλου του αραβικού κόσμου. Η μη η μη δυνατότητα πρόθεση τη συνευτική διαδικασία περιπλέκει όλα τα άλλα περιφερειακά προβλήματα. Όλα αυτά τα θέματα απαιτούν συνεργασία στενή μεταξύ των χωρών τη ε, Συμβουλίου του Κόλπου και τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ταυτόχρονα όμω οι χώρε του κόλπου οι ίδιε θέλουν να διευρύνουν τι διεθνεί του σχέσει και είναι έτοιμε ενεργά να προωθήσουν ε, τα εθνικά του συμφέροντα. Περισσότερο από ό,τι κατά παρελθόν η Ευρώπη δεν είναι ο αποκλειστικό εταίρο λόγω ιστορικών δεσμών με την περιοχή. Ανταυτού η Ασία, η Αφρική και ακόμα και η Λατινική Αμερική θα διδραματίσουν κάποιο ρόλο οικονομικό και πολιτικό στην περιοχή. Τώρα θα στραφώ στο δεύτερο ερώτημα, γιατί θα πρέπει οι χώρε του Συμβουλίου του Κόλπου να είναι μια βάση για μια αναζωογονημένη εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώση και των χωρών αυτών. Ε, λοιπόν, αυτέ οι χώρε είναι σημαντικέ γεωπολιτικώ και έχουν μεγαλύτερη επιρροή στον αφορά τι εξελίξει στην περιοχή. Όπω ανέφερε μια έκθεση πρόσφατα, λέει ότι οι χώρες του κόλπου ηγούνται, επηρεάζουν τις εξελίξεις, έχουν μεγαλύτερες οικονομικές ευθύνες, ε, ε, δείχνουν ότι έχουν οικονομική και κοινωνική εμπιστοσύνη και ε, αποκτούν επίγνωση της νέας θέσης που αποκτούν σαν περιφερειακή δύναμη που ξεπερνά τις υπόλοιπες αραβικές χώρες. Η στην Βουλή του Κόλπου ε, θέλουν να υποστηρίξουν την πολιτική σταθερότητα, έχουν σωστή ε, μετριοπαθή ιδεολογία, έχουν οικονομικό δυναμισμό και θέλουν να προχωρήσουν με προγράμματα περιφερειακής ολοκλήρωσης. Λοιπόν, θα πρέπει να ειδωθεί βασική λοιπόν αυτή η σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτέ τι χώρε. Υπάρχουν διάφορε στοιχεία που αφορούν αυτή τη σχέση. Οι χώρε ε, του, του, κόλπου ε, εξακολουθούν να αλλάζουν σημαντικά και γίνονται οικονομικέ και πολιτικέ μεταρρυθμίσει σε κάθε χώρα και από την ίδια την εμπειρία τη η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει τι διαδικασίε μέσω υπευθύνων και μετρημένων πολιτικών. Οι χώρε του Συμβουλίου του Κόλπου ήταν στην πρώτη γραμμή όσον αφορά ε, την προμήθεια στον υπόλοιπο κόσμο φτηνής και αξιόπιστης ενέργειας, αξιόπιστη φωτισμού ενέργεια και παραμένουν σταθεροποιητική δύναμη όσον αφορά την αγορά πετρελαίου. Και είναι, οριμάζουν οι χώρε αυτέ και συμβάλλουν στην περιφερειακή σταθερότητα και συμβάλλουν στι προσπάθειε ειρήνευση μέσω ε, διαμεσολάβηση διπλωματική και επιλύσεω σειράξεων, όπω ειρηνευτική, η αραβική ειρηνευτική ε, πρωτοβουλία για να σταματήσει η σύραξη μεταξύ Αραβών και Ισραηλινών ε, είναι κάτι που υπευλήθη από τη Σαουδική Αραβία και με συμμετοχή της Παλαιστίνης, του Ιράκ, του Λιβάνου, της Ιεμένης και του Σουδάν. Μάλλον στην Παλαιστίνη, στο Ιράκ, στο Λίβανο, στην Ιεμένη Σουδάν. Λοιπόν, όλε αυτέ τι προσπάθειε δείχνουν ότι θα είναι καλό να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την περιοχή και τελικά οι χώρε του Συμβουλίου του Κόλπου έχουν προχωρήσει όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση. Οι πρόσφατε συζητήσει οδήγησαν σε καλύτερη συντονισμένη προσέγγιση και είχαν σαν αποτέλεσμα συγκεκριμένα συγκεκριμένου στόχου όπω Τελωνιακή Ένωση, σχέδια για μια κοινή αγορά και θέλουν και ένα κοινό νόμισμα και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα όπω ένα συνδρομικό δίκτυο και ένα δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια. Μέσω τη συμμετοχή του, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στην περιφερειακή αυτή προσπάθεια. Έχοντα όλα αυτά υπόψη, Βλέπουμε ότι χρειάζεται μια πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω βάσει κοινών συμφερόντων. Θέλουμε σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή και ισχυρού πολιτικού δεσμού. Αν βάλουμε και πολιτική συνισταμένη στην... στι σχέσει αυτέ, αυτό είναι κάτι σημαντικό, διότι έχουν σημασία αυτέ οι χώρε. Και οι, οι χώρε δίνουν σημασία σε αυτό το θέμα. Τι θέλουν περισσότερο, να έχουν σοβαρού συνομιλητέ. Να θεωρηθούν ότι μπορούν να βοηθήσουν να συμβάλλουν σε επίλυση διαφόρων προβλημάτων και στην βελτίωση τη ασφαλεία στην περιοχή θέλουν να συμμετέχουν, όχι να τους λένε τι να κάνουν. Θέλουν να γίνονται σεβαστά τα εθνικά τους συμφέροντα και να μην θεωρούνται ότι είναι απλώς καταναλωτές και ότι πληρώνουν για διάφορους επιτυχιαφόρων στόχους. Τώρα τελικά θέλω να στραφώ στο τελευταίο ερώτημα και να κάνω συγκεκριμένε προτάσει. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω με τι χώρε αυτέ. Πέρα από την Υπουργική Σύνοδο ε, που συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, που λαμβάνει μια χώρα μία φορά το χρόνο, θα πρέπει να γίνεται δύο φορέ Σύνοδο Κορυφή και αυτή θα είναι αυτό θα είναι σωστό μήνυμα στην περιοχή ότι λαμβάνουμε σοβαρά αυτή τη σχέση. Θα πρέπει να κάνουμε μια δήλωση πολιτική για τι χώρε του κόλπου Όπω είδαμε και με τη Μέση Ανατολή και τη σχέση με τη Μεσόγειο και την εταιρική σχέση λαμβάνοντα υπόψη τη προσεγγίσει ακολουθούμε για άλλε περιοχέ του κόσμου δεν ξέρει αυτή η περιοχή Πού στέκεται, θα το διορθώσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ε, από ε, τι δύο πλευρέ πολιτικό-στρατηγικό διάλογο. Θα επιτρέψει καλύτερο συντονισμό των πολιτικών και να αποφεληθούμε και από τις δεσμούς που έχουν οι χώρε στο Συμβουλίου του Κόλπου με διάφορες χώρες που είναι προβληματικές στην περιοχή. Θα πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει αντιπροσώπηση, εκπροσώπηση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στι χώρε αυτέ. Δεν αρκεί η εκπροσώπηση σημερινή για να αντιμετωπίσει ε, σωστά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή του Κόλπου. Χρειάζεται μια αυξημένη παρουσία στις Ευρωπαϊκές Ενώσεω. Θα πρέπει να αυξηθεί, αυξηθούν οι δραστηριότητε διπλωματία τη Ευρωπαϊκής Ενώσης στην περιοχή. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νομίζω ότι παρόμοιε στο στο παρελθόν ήταν άκρο επωφελή. Και συνεχίζονται οι προσπάθειε. Δεν σταματά αυτή η προσπάθεια. Τέλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε του κόλπου θα πρέπει να εξοντενήσουν τι πολιτικέ όσον αφορά το Αφγανιστάν, την Ιεμένη και το Πακιστάν. Αυτέ οι γειτονικέ χώρε του κόλπου είναι κρισίμου σημασία στη σταθερότητα των χωρών του Συμβουλίου του κόλπου και για την Ευρώπη. Η βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω συνήθω έχει πολλού όρου που ε, τίθενται ε, και λοιπόν σε τοπικό επίπεδο υπάρχει αντίσταση γι' αυτό. Δοθέντως ότι οι χώρες του Συμβουλίου της, ε, του κόλπου ε, ε, βλέπονται πιο καλό μάτι τι χώρε τη περιοχή, θα μπορούσαν να εφαρμόσουμε σωστό επιμερισμό των προσπαθειών σε προσπάθειε συνεργασία όσον αφορά τη βοήθεια που χορηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε του κόλπου. Θα πρέπει να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν ε, χάσαν πολλές ευκαιρίες, δεν έχει κλείσει όμως η πόρτα, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Θα πρέπει οι σχέσεις να έχουν το σωστό πολιτικό πλαίσιο και αυτές οι δυνατότητες θα μπορούν τελικά να μετατραπούν σε πραγματικά επιτεύγματα. Σε πρόσφατη έκθεση που είδαμε πρόσφατα δημοσιεύεται, είπε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να βασιστεί στι μετριοπαθεί ε, πολιτικέ των χωρών του Συμβουλίου του Κόλπου για να προωθηθεί ένα πρόγραμμα τη περιοχή που βασίζεται στι δικέ τη επιταγέ για πολυμερή προσέγγιση. Θα πρέπει οι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να προωθηθούν όσον αφορά διαχείριση των συγκρούσεων, την πρόθεση τη ειρήνη και θα πρέπει να απογραμμίζεται και η αρχή τη κοινή κυριαρχία. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή ε, πολιτική στον κόλπο να ξεκινήσει από τη συνεργασία της με τις χώρες του Συμβουλίου της, ε, του κόλπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόκ. Και τώρα ο κύριος Ρουζιέ Φιλίπ Μπερτότσι έχει το λόγο. Παρακαλώ, αν μπορέσετε να τηρήσετε το χρονικό όριο των 10 λεπτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιδέες ε, που συνέλεξα από 15 ετή πείρα σε διάφορους τομείς των σχέσεων με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου ζήτημα που θα μπορούσαμε να σημειώσουμε είναι ότι την τελευταία 20 ετία σχεδόν αποκλειστικό επίκεντρο των ε, διαπραγματεύσεων ελευθέρου εμπορίου ήταν μια μαύρη τρύπα που απορρόφησε όλη την ενέργεια που κανονικά θα μπορούσε να είχε αφιερωθεί και σε άλλους στρατηγικούς τομείς αυτής πολύ σημαντικής αλλά δυστυχώς παραμελημένης σχέσης. Εν τω μεταξύ ο κόλπος ε, ε, και η περιοχή του κόλπου έχει εξελιχθεί όχι μόνο ραγδαία αλλά και προς διάφορες κατευθύνσεις που δεν έγιναν ε, δεόντως αντιληπτές πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι σαν φουτουριστικός κόμβος η περιοχή του κόλπου, βρήθη οικονομικής και κοινωνικής ευρηματικότητας και είναι ένα εργαστήριο πολυεθνικών, πολυσύνθετων κοινωνιών που θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και επίσης έχει τεράστια ε, επίδραση μέσω διάφορων ανθρωπιστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων προ διάφορε περιοχέ του κόσμου. Ενδιαφέρουσα είναι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και στην ε, Μέση Ανατολή και στην ε, Ασία, αλλά και στην Ινδία, στο Ιράν και στην Ανατολική Ασία. Είναι πολλέ οι επιρροέ που δέχεται η περιοχή του κόλπου. Αν λοιπόν ε, δεν ε, επιλεχθεί το σωστό επίπεδο στρατηγικής διπλωματίας με το ε, Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόσμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της θα στερηθεί τεράστιο δυναμικό πόρο ενός πολύ ζωτικού εταίρου, ενός νευραλγικού εταίρου σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας, οικονομικής ανάπτυξης, τεχνολογίας και έρευνας και καινοτομίας. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που κατά τη γνώμη μου ε, δείχνει τι θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει αν είχαμε ασχοληθεί και με άλλα θέματα εκτός από τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πασχίζει να φτάσει στο 3% κατόφλι του ΑΕΠ για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Και παρόλο που έχουμε ηγετικό ρόλο, αρχίζουμε και μένουμε πίσω ως προς την Κίνα που έχει δύο εκατομμύρια ερευνητές το χρόνο, την Ινδία που κάθε χρόνο παράγει τεράστιο ρυθμό μηχανικών και μάλιστα πέρυσι ε, οι 2.000 ε, και με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανανοτεχνολογία, η Ινδία επίσης εντυπωσιακό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Όλες αυτές οι χώρες έχουν ε, ξεκινήσει πολύ φιλόδοξα προγράμματα ε, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας. Είναι ανοησία λοιπόν ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει ήδη εγκαινιάσει όχι μόνο στρατηγική συνεργασία με τις χώρες του Συμβουλίου συνεργασία του Κόλπου για θέματα επιστημονικής έρευνας, για τεχνολογία αλλά και χρηματοδότηση στρατηγικών βιομηχανιών αλλά και σε ό,τι αφορά τα δημόσια ταμεία πλούτου, τα sovereign wealth funds που έχουν ρευστότητα τρισεκατομμυρίων στον κόλπο και μερικά τέτοια κονδύλια ψάχνουν να επενδύσουν σε νευραλγικές τεχνολογίες που θα είναι σημαντικές για τον 21ο αιώνα, όπως θα είναι η ρομποτική, η νανοτεχνολογία, ε, καθαρής ενέργειας, ε, υδρογόνου. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να έχουμε όλο και πιο πλούσια συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χρηματοδότησης τέτοιων ε, δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της χρηματοδότησης ε, των δημόσιων ταμείων πλούτου, των sovereign wealth funds, γιατί έχουν τεράστιο δυναμικό, τεράστια ρευστότητα, οπότε είναι προ όφελο τη Ευρωπαϊκής Ένωση να ξεκινήσει τέτοια συνεργασία. Και αντί να προσπαθήσει να ευθυγραμμιστεί με την Ινδία, την Κίνα, την Κορέα, τις αναδυόμενες ε, τεχνολογικές δυνάμεις, καλό θα ήταν ε, να επενδύσει και στη συνεργασία, στρατηγική συνεργασία με τις χώρες ε, Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Και αν εξετάσουμε όλα τα γνωστά στοιχεία που καθιστούν τόσο απαραίτητες τις σχέσεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις είναι να προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια φιλόδοξη πρόταση, ένα φιλόδοξο όραμα και να προτείνει μια στρατηγική συνεργασία εταιρική σχέση προς το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Γιατί αν εξετάσουμε τις πολιτικές δομές αλλά και άλλους τομεί που δεν ε, έχουν ακόμη οριμάσει, σε τελική ανάλυση μόνο με ένα τέτοιο φιλόδοξο όραμα, μόνο με μια τέτοια πρόταση και συζήτηση με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου μπορούμε ε, να αρχίσουμε να του δίνουμε σάρκα και ωστά. Γιατί το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου δεν, περιλα... δεν περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο κατάλογο για ανταλλαγή εμπειριών, ε, εμπειρογνωμόνων, και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα ήδη έγιναν. Αυτό που περιμένει το Συμβούλιο Συνεργασία του Κόλπου είναι μια γνήσια στρατηγική πολιτική και περιμένει να γίνει ισότιμο εταίρο Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια τέτοια στρατηγική συνεργασία. Οπότε τέτοιου είδου πρωτοβουλίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδιαίτερα με τις ενισχυμένες αρμοδιότητες που έχει από τη συνθήκη της Λισαβόνας για τις εξωτερικές σχέσεις και για τις εμπορικές συμφωνίες, είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μετά το τελευταίο Συμβούλιο του Λουξεμβούργου που έδωσε μια νέα όθηση. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στα χέρια του μια ιστορική ευκαιρία, γιατί μπορεί πια να αποφασίσει να καταρτήσει δύο ακόμη ψηφίσματα και να εκπονήσει δύο ακόμη εκθέσεις, αλλά μπορεί να αποφασίσει να προτείνει και κάτι παραπάνω, που θα ήταν μια στρατηγική, συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης πολυεπίπεδη που θα περιλαμβάνει όλε τι διαστάσει τη σχέση με το Συμβούλιο συνεργασία του Κόλπου και θα προβλέπει την απαραίτητη κατάρτιση, προσωπικό και χρηματοδότηση καθώ και τι δομέ για να υλοποιηθεί αυτή η συνεργασία. Γιατί φυσικά θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτή τη σχέση, θέλουμε να βελτιώσουμε την παρουσία και τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και αν δεν είμαστε έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε μια τέτοια αναβάθμιση της παρουσίας δεν πρόκειται να την υλοποιήσουμε. Έχουμε 172 εκατομμύρια, αλλά είναι, είναι ψυχία, αμεληταίο ποσό σε σχέση με αυτά που θα χρειάζονται για να επενδύσουμε σε μια νέα στρατηγική σχέση στην περιοχή του κόλπου. Επειδή όμως υπάρχει, έχει δοθεί νέα όθηση, χάρη στο κοινό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και χάρη στις ε, δυνατότητες που υπάρχουν είτε να εμείνουμε στην ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών είτε να μην ε, συγκεντρώσουμε όλη την ενέργεια των διαπραγματεύσεων σε αυτή τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, θα ήταν σκόπιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανάλογα με την έκβαση των ψηφισμάτων και των συζητήσεων, να χρησιμοποιήσει την επόμενη, το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει το 2011 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα που θα διαμορφωθεί μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβουλίου Συνεργασία του Κόλπου, ώστε να προβάλλει στη δημόσια συζήτηση τα ψηφίσματα αυτά. Και νομίζω ότι τρία θα ήταν τα πλεονεκτήματα. Καταρχήν, θα εξασφαλίσετε την ε, παρουσία ε, υψηλόβαθμων και ηθινόντων στην παρουσίαση αυτή. Οπότε θα δώσετε μια μεγαλύτερη προβολή και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και πολιτική προβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της αξίας του κοινοβουλευτισμού και της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει το παρόν ως θεσμική οντότητα γιατί θα εκπροσωπείται από συνεργασία ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Θα είναι τρισυπόστατη εκεί η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σίγουρα η συζήτηση των ψηφισμάτων θα γίνει και με προσώπους επιχειρηματικών κύκλων και της οικονομικής κοινότητα ε, του Συμβουλίου Συνεργασία του Κόλπου και αυτή θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να δοθεί ένα πρόσωπο σε αυτή την θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρώπης που θα μπορούσε να είναι και παράδειγμα προς μίμηση για πολλές περιοχές του κόσμου αλλά ταυτόχρονα θα ήταν ε, και το καλύτερο παράδειγμα και καλύτερη προβολή, γιατί επιτέλου θα δουν οι κάτοικοι του κόλπου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προτείνει κάτι καινούργιο και είναι δεσμευμένη και πρόθυμη να περάσει σε μια νέα εποχή, προβλέποντας τι κατάλληλε δομές, προσωπικό, χρηματοδότηση, πόρους για μια τέτοια νέα συνεργασία. Οπότε μια τέτοια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είχε πραγματικά ιστορική σημασία και θα συμβάλλει στο να αναβαθμιστεί η συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόσμου που πραγματικά ο πολυεπίπεδος ε, κόσμος παγκοσμιοποιημένος με τις πολλές προκλήσεις καθιστά απαραίτητη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπερτότσε για κάποιος, κάποια σχόλια, κάποιες ερωτήσεις θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο Ντομινίκ Μποντής. Στον κύριο Ντομινίκ Μποντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Μπερτότσι και στον κύριο Κοχ. Οι αναλύσεις τους είναι πολύ χρήσιμες για την Επιτροπή μας ε, κατά την εκπόνηση της έκθεσής μου. Θα ήθελα να πω ότι η πρέσβυρα της, ε, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, η κυρία Αμάλε Λαμάντ, που είναι παρούσα στην αίθουσα, αλλά και η πρέσβυρα του, του Κουβέιτ, κυρία Μαντήρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το Κουβέιτ αυτή τη στιγμή προεδρεύει στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και οι δύο κυρίες είναι παρούσες στην αίθουσα. Θα υποβάλω σύντομα τις ερωτήσεις μου για να έχουμε χρόνο για τις απαντήσεις. Αναφέρθηκε εκτενώς το θέμα αναβάθμισης των σχέσεων των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόσμου υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε όμως να μας πείτε πώς ε, οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, οι Αραβικέ χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, πώς βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς την αντιλαμβάνονται και τι προσδοκούν από αυτήν. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Πολύ σωστά και εύστοχα επισημάνατε το θέμα της ασφάλειας ε, στην περιοχή που είναι πολύ ανησυχητικό γιατί έχουμε τον πόλεμο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Εκεί έχει μειωθεί η αξιοπιστία των Αμερικανών σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να ρυθμίσουν δια της βίας μια περιφερειακή κατάσταση. Το Ιράν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση και να ε, ενισχύσει τη θέση του με διάφορες έρευνες που κάνει στα θέματα του πυρηνικού εξοπλισμού, κάτι που είναι ανησυχητικό και για τις ε, χώρες του κόλπου, γιατί μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο μιας σύγκρισης και να γίνουν τα παράπλευρα θύματα μιας τέτοιας σύγκρουσης. Απόδειξη, ένα συμβόλαιο οπλισμού, ρεκόρ μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, που υπογράφει την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι που δείχνει ότι συμπαρασύρεται η ευρύτερη περιοχή σε μια κούρσα εξοπλισμών. Επίσης ε, αναφέρατε μια αναπτυσσόμενη διπλωματία των, των αραβικών χωρών του, κόσμου, του κόλπου. Μπορούμε να μιλήσουμε όμως για μια ομοιόμορφη, ομοιογενή, συγκλίνουσα διπλωματία. Όταν βλέπουμε το χάσμα που χωρίζει μερικές φορές ε, την ε, Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, από το Εμμυράτο του Κατάρ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε Μποντής. Ο, Μάριο, ο κύριος Μάριο Νταβίδ που είναι εισηγητής για σύνταξη γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ντομινίκ Μποντής γιατί ανέφερε την έκθεση σας ευχαριστώ θερμά. Άλλωστε αυτές τις δύο εκθέσεις ανέφεραν και οι δύο προσκεκλημένοι μας. Οι σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου είναι πολύ δυστυχώς χαλαρές, πολύ ασθενείς και στερούν ε, κατά πολύ σε σχέση με τις προσδοκίες μας. Το απόγευμα γύρω στις 5 θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στην οποία συμμετέχω και θα γίνει μια πρώτη συζήτηση επί της εκθέσεως. Αλλά τώρα μια και βρισκόμαστε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα ήθελα να σας υποβάλω μια ερώτηση και να κάνω και μια πρόταση προς τον Ντομινί για την έκθεσή του γιατί αφορά το πολιτικό σκέλος και όχι το εμπορικό. Νομίζω ότι σκόπιμο θα ήταν για να δώσουμε ένα μήνυμα του ενδιαφέροντος Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την περιοχή αυτή του κόλπου. Ε, ήταν μία πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, διεξαγωγή της διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Βέβαια αρχίζει και γεμίζει υπερβολικά το χρονοδιάγραμμα των Συμβουλίων Κορυφής. Καλό θα ήταν όμως σε αυτή την πλούσια ατζέντα συμβουλίων κορυφής να προσθέσουμε ακόμη ένα αυτό με το Συμβούλιο Συνεργασία του Κόλπου και να ε, διοργανώνουμε ετησίω τέτοιο είδου Συμβουλίο κορυφή. Κάτι άλλο που θα μας ενδιέφερε είναι να δούμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης πώς θα απαντήσουμε στο ερώτημα που μας έδωσε ο δόκτωρας Κοχ δεν υπάρχει μία μόνιμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ε, έξι χώρες ε, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Σας ευχαριστώ κύριε Νταβίτ. Κυρία Νίμπλερ, πρόεδρος της αντιπροσωπείας σχέσεων με τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στις εργασίες της Επιτροπής σας σήμερα. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι, να καταρχάς να πω ότι ε, θεωρώ την εξαιρετική πρωτοβουλία της Επιτροπής σας για την ε, έκθεση αυτή, για τη συνεργασία με τις χώρες του κόλπου και νομίζω ότι αυτό τονίζει την πτυχή της συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο, όχι μόνο από στρατηγικής άποψης, αλλά και σε πρακτική εφαρμογή να προσπαθήσουμε να συνεργαζόμαστε με τις ε, χώρες για να έχουμε πολιτικά ε, ωφέλη. Θα ήθελα δύο συγκεκριμένα στοιχεία να θίξω. Η αντιπροσωπεία μου πριν από κάποιους μήνες μετέβη στο Κατάρ και στο Κουβέιτ και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, επικεφαλής ε, του Κουβέιτ και της ε, συνεργασίας και των χρόνων συνεργασίας. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η υποδοχή μας και εξαιρετική συνεργασία μας, οι συζητήσεις μας. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι είναι εξαιρετικά άσχημη η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Αν θα μπορούσατε λοιπόν να το σχολιάσετε και εσείς αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο στο ΡΙΑΔ ε, εκπροσωπείται σήμερα. Και θα ήθελα και στα πλαίσια της έκθεσης αυτής να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα πλαίσια της διεύρυνσης ε, της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάφορες υπηρεσίες. Να την καλέσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει τι μπορεί να γίνει για την εκπροσώπηση στις περιοχές αυτές. Θα πρέπει να είναι ορατή η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο ένα γραφείο στο ΡΙΑΤ, θα πρέπει να υπάρχει ε, δική μας εκπροσώπηση και σε άλλα κράτη. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι θα πρέπει να διαφημίσουμε αυτό που προσφέρουμε και ως Ευρωπαίοι. Είμαι εισηγήτρια και για την Επιτροπή Βιομηχανίας για την ε, έκθεση αυτή. Και διαπιστώσαμε στις συζητήσεις μας με το Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, στο Κατάρ, ότι τα προγράμματα ερευνητικά που διαθέτουμε, το Erasmus Mundus, για παράδειγμα, αυτά που προσφέρουμε στις φοιτητέ της περιοχής δεν είναι καθόλου γνωστά. Μία έκκληση λοιπόν απευθύνω για τον ίδιο μας τον εαυτό να φροντίσουμε τα προγράμματα συνεργασίας να ανοίξουν και να διαφημιστούν στην περιοχή. Να πούμε ότι καλούμε για παράδειγμα τους νέους ανθρώπους να έρθουν στην Ευρώπη. Να το διαφημίσουμε. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις. Μάλιστα, επί σειρά ετών διαπραγματευόμαστε τις εμπορικές συμφωνίες και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, αλλά σημαντικό είναι να αναλύσουμε στην περιοχή του κόλπου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε η κοινή στόχη. Στην ενέργεια, στην οικονομική συνεργασία, στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Θα πρέπει τα κοινά συμφέροντά μας να τα βάλουμε κάτω και με μικρά βήματα να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Φυσικά θα πρέπει να διατηρήσουμε θα, πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανά το όραμα της ε, συμφωνίας FTA και της υπογραφής της συμφωνίας, αλλά ας προχωρήσει η επιτέλους και η συνεργασία μας με τους εταίρους μας από τις χώρες του κόλπου. Σε ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ. Στις 4 προβλέπεται συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας. Έχουμε λίγο χρόνο λοιπόν για ερωτήσεις και παρακαλώ να τις συγκεντρώσετε ερωτήσεις σε ένα λεπτό ή δυνατόν. Όσον αφορά τα σχόλια θα υπάρξουν και άλλες περιστάσεις πριν από την έγκριση των εκθέσεων των συναδέλφων. Θα συζητήσουμε αυτά. Ο κύριος Άτκινς ένα λεπτό, ένα ερώτημα αν έχετε την καλοσύνη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξυπακούεται ότι η συνεργασία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου είναι κάτι που όλοι εγκρίνουμε. Όπως θα έλεγαν οι Αμερικανοί, εδώ είναι ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, θα πρέπει να εξετάσουμε ε, τα θεμελιώδη θέματα της συγκρούσεως στη Μέση Ανατολή ευρύτερα, όχι μόνο μεταξύ των ε, Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Ερωτήσεις. Το Συμβούλιο συνεργασία του Κόλπου τι κάνει για να αντιμετωπίσει τι διεθνεί εντάσει που υπάρχουν. Δεύτερον, είστε ενωμένοι σαν χώρε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τρίτον, τι κάνετε για να πιέσετε τι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτω ώστε να ακολουθεί ισότιμη προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τις διαφορές που υπάρχουν. Τέλος, ένα θέμα που προβληματίζει και εδώ στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μετράει πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά. Τι συγκεκριμένο μπορούμε να κάνουμε και εμείς και εσείς, ούτω ώστε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει αξία και να έχει αποτελέσματα. Κυρία Άτκιν, συγχαρητήρια. Καταφέρατε να κάνετε τέσσερις ερωτήσεις ένα λεπτό. Φόξ, ένα λεπτό για μία ερώτηση σας παρακαλώ. Κύριος Φόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Είπατε ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε μια πιο στενή σχέση με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, να μην εστιαστούμε μόνο στο εμπόριο. Ποια ήταν η αντίδρασή τους όμως στην ανάγκη δια δογματικού, διαθρησκευτικού, αν θέλετε, διαλόγου. Και κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εμβάθυνση των σχέσεων σε άσχετου τομεί πέρα από το εμπόριο, που δεν συνδέονται άμεσα με το εμπόριο. Σα ευχαριστώ κύριε Φόξ. Μέχρι τι 4 θα πρέπει να υποδιαρέσετε το χρόνο ανάλογα για να δώσετε απαντήσει. Και να απαντήσετε στα θέματα που θεωρείτε τα πιο επίκαιρα για να απαντήσετε. Έχετε το λόγο κύριε Κόχ. Ευχαριστώ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις που θέσατε. Να ξεκινήσω από το πρώτο, γιατί νομίζω ότι σχετίζεται με πολλά άλλα θέματα που αναφέρθηκαν και το πώς θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η θεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόλπο. Όπως είπατε δεν είναι ιδιαίτερα ορατή και αυτό σχετίζεται ιδιαίτερα με το γεγονός ότι υπάρχει για παράδειγμα μόνο ένα γραφείο στο Ριάντα και ο πρεσβευτής εκεί είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά ένας είναι μόνος του. Τι να κάνει, πώς να καλύψει έξι κράτη. Και όπως είπα και εισαγωγικά, οι πολιτικές σχέσεις, οι άμεσες πολιτικές σχέσεις είναι απαραίτητες, απόλυτα απαραίτητες στην περιοχή του κόλπου. Αν θέλει κανείς να τον πάρουν στα σοβαρά πρέπει να είναι εκεί. Να μιλάει με τους πολιτικούς αρχηγούς και το να το κάνει τώρα ένα άτομο για έξι χώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτη στην περιοχή αυτή και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Και επίσης Πολλές από τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, περνάνε μέσα από το πρίσμα του FTA. Ο κόσμος δηλαδή τι λέει. Ε, αν δεν καταφέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψει τη συμφωνία αυτή ε, ζώνης ελευθερίου εμπορίου, πώς να την πάρουμε στα σοβαρά και άλλα θέματα. Άρα, είναι δύσκολο να διαδώσουμε το μήνυμά μας. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχουν πιο πολλοί πιο πολλά πιο πολλή διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο έντονη η διαβίβαση του μηνύματος που θέλουμε να δώσουμε, μεγαλύτερες επαφές με την πολιτική ηγεσία. Να υπάρχει, για παράδειγμα, ε, ετήσια ή κάθε δύο χρόνια μια σύνοδος. Αν υπάρχουν οι καλές πολιτικές σχέσεις σε ανώτερο επίπεδο, αυτό θα ανοίξει τις πόρτες σε πολλούς άλλους τομείς σε ό,τι αφορά τη διπλωματία τώρα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια νέα περιοχή. Με το Ιράκ κατέστη σαφές ότι ακόμα χρειάζονταν οι χώρες του κόλπου της είπα για προστασία, για στρατιωτική προστασία. Αλλά οι είπα δεν εντρούν απαραίτητα πάντα υπέρ ε, του συμφέροντος των χωρών του κόλπου. Πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθεί. Μετά το επεισόδιο με το Ιράκ υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση, δίδεται μεγαλύτερη, έμφαση από πλευρά των χωρών του κόλπου να δραστηριοποιηθούμε πιο πολύ και οι προσπάθειες διαμεσολάβησης ε, γίνονται σε πολλές ε, περιπτώσεις. Ακόμα και για να κρατηθεί ανοιχτή, αν θέλετε, και η πόρτα και με το Ιράν. Γιατί εντάξει μπορούν να συμφωνούν οι χώρες ε, του κόλπου ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα από πλευρά του Ιράν, αλλά χρειάζεται να έχουν συνομιλίες, να έχουν σχέσεις με το Ιράν. Για παράδειγμα το Ομάν. Κανείς δεν θέλει στην περιοχή εκείνη να κάνει το Ιράν εχθρό του, γιατί στη τελική ανάλυση δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφική πραγματικότητα και το Συμβούλιο συνεργασία του Κόλπου αναγκαστικά θα έχει πάντα σχέση με το Ιράν. Άρα συνολικά πρέπει να πω ότι υπάρχει μία α, κοινή θέση, υπάρχει μία κοινή αντίληψη για το ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πώ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και πάντα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα επιμέρους θέματα αλλά επί της αρχής υπάρχει κοινή, επικρατεί κοινή αντίληψη και υπάρχει μια κοινή θέση για τα προβλήματα στην περιοχή. Αυτά τα δύο θέματα ήθελα βασικά να αναφέρω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κόχ. Κύριο Μπερτότσι έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα το πώς γίνεται αντιληπτή η Ευρώπη από τις χώρες του κόλπου, έχω να το εξής. Οι διαπραγματεύσει για τη Συμφωνία Ελευθέρων Διαπραγματεύσεων είναι σαν ένα πέπλο που κάλυψε όλα τα άλλα θέματα. Απ' την άλλη πλευρά δεν υπήρξε κανένα πρόγραμμα ή χρήματα που διατέθηκαν για ενεργή πρόθεση της Ευρώπης και προβολή της Ευρώπης στον κόλπο. Είμαστε ακόμα δύο άγνωστα σύμπαντα εμείς και οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Η Ευρώπη, ίσως για λόγους πολιτισμικούς, δεν θέλει να προβάλλει την εικόνα της υπερδύναμης. Προβάλλει μια ήπια δύναμη. Δεν ξέρω γιατί η Ευρώπη δέχεται την ε, ίδια την ιδέα της δικής της ε, πτώσης, αν θέλετε. Και εκεί όλα γίνονται αντιληπτά ως θέματα ισχύω. Αν δεν γίνεις αντιληπτός ως ισχυρός, ως ισχύς, δεν σε, δεν σε ακούν. Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου θέλει την Ευρώπη ισχυρή. Διότι ξέρει ότι έχει τρόπους να χρησιμοποιήσει ε, τη δύναμή της ε, για να προωθήσει την ειρήνη, την πρόοδο και την συνεργασία. Και αυτό ταιριάζει και ιστορικά με τη διπλωματία ε, των χωρών του κόλπου. Ήταν πάντα φιλιρινικές, ήταν αδέσμευτες, έδιναν τα μεγαλύτερα ποσά ως βοήθεια στον κόσμο Άρα υπάρχει μεγάλη δυνατότητα διπλωματικής σύγκλησης, αλλά ο κόλπος θέλει να αισθανθεί ότι η Ευρώπη είναι ισχυρός φορέας. Όχι μόνο να βοηθήσει την ολοκλήρωση των ενευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Πρέπει να δοθεί ισχύς, δύναμη στη σχέση. Συμφωνώ με το έγγραφο που κυκλοφόρησε. Δηλαδή, μια ετήσια σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρών του κόλπου είναι κάτι απαραίτητο, όχι επειδή είναι της μόδας. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν πάρα πολλοί πολυμερείς μεγάλου εύρου συζητήσεις. Καμιά φορά πιο, μικρά, πιο μικροί σχηματισμοί είναι πιο αποτελεσματική. Είναι θέμα ανοτροπίας, ψυχολογίας, πολιτισμικό θέμα. Το πώς οι πολίτες του κόλπου βασίζουν τις σχέσεις τους σε εμπιστοσύνη σε προσωπικές σχέσεις, σε προσωπικό επίπεδο. Και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης θα πρέπει να επενδύσουν χρόνο για να δημιουργήσουν ισχυρές προσωπικές σχέσεις με τους ηγέτες των ε, χωρών της, ε, του κόλπου και με, τους, ε, με την ελίτ την κοινωνική και την επιχειρηματική. Μια σύνοδος κορυφής ετήσια θα δώσει σάρκα και οστά στη σχέση. Δεν θα συζητούνται μόνο πολιτικά διπλωματικά θέματα. Η δομή της εξουσίας και η διοργάνωση των κυβερνήσεων και των χωρών στις χώρες του Συμβουλίου του Κόλπου ακολουθούν μια πυραμιδική ε, ε, ιεραρχία και χρειάζεται συζήτηση των βασικών θεμάτων. Θα βγαίνουν προσανατολισμοί από τις συνόδους κορυφής έτσι. και τελικά οι αποφάσεις θα έχουν αποτελέσματα. Τώρα για το διαπολιτισμικό διάλογο και για το διαθρησκευτικό διάλογο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τίνουμε πάντα να βλέπουμε με άλλο τρόπο αυτό το διαθρησκευτικό διάλογο. Πώς οι Ισλαμικές χώρες βλέπουν, παραδείγματος χάρη, τα σκεφτικά θέματα και το σκεφτικό διάλογο. Η Ευρώπη σωστά υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι χριστιανικές της ρίζες. Όμως, πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δεχτεί πλήρως το ότι έχει χριστιανική κληρονομιά, έχει εβραϊκή κληρονομιά, μουσουλμανική κληρονομιά ε, η Ευρώπη. Θα πρέπει να δεχτεί η Ευρώπη ότι το Ισλάμ είναι στην Ευρώπη από παλιά. και συνέβαλε τα μάλα στον πολιτισμό της Ευρώπης σε διάφορα επίπεδα. Και σήμερα η Ευρώπη είναι μια μουσουλμανική ήπειρος. Αύριο μάλλον θα είναι. Θα έχουμε 38 εκατομμύρια μουσουλμάνους που θα ζουν στην Ευρώπη μέχρι το 2020-2025. Είναι περίπου όσο είναι ο πληθυσμό των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Θα πρέπει να δεχτούμε ότι η Ευρώπη είναι επίσης και Ισλαμική Ήπειρος και από αυτή την έποψη ο διάλογος μπορεί να λάβει μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Μπορεί να γίνει συζήτηση επί της ουσίας και όχι μόνο επί αντιλήψεων και θεωριών. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα τους πολιτισμικούς και ιστορικούς δεσμούς και μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο βάσει ουσίας και όχι βάσει παρεξηγήσεων και λανθασμένων αντιλήψεων. ανήκουμε όχι μόνο σε κοινή ιστορία όπως σας είπα, έχουμε ρίζες από τον Αβραάμ, αλλά ανήκουμε και σε ένα γεωγραφικό σύνολο. Ρωσία, Τουρκία, Ευρώπη, Μαγκρέμπ, Μασρέκ, Κόλπο. Και σε όλη αυτή τη μεγάλη περιοχή υπάρχουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί, ταυτόχρονα τίνουμε να δημιουργούμε μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου που θα είναι μεγαλύτερη στον κόσμο που συμπεριλαμβάνει όλες τις μεσογειακές χώρες, τον κόλπο, την Ευρώπη. Η Τουρκία ήδη είχε τελειωνιακή ένωση, ίσως κάποια μέρα ε, θα προδέσει τη σχέση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια, ένα τεράστιο μόρφωμα γεωγραφικό που είχε, είχε πάντα λογική Ευρασία, Ρωσία, Τουρκία, ε, ε, Ευρώπη, κόλπος, Μασρέκ, Μαγκρέπ, πάντα για τους αυτού που ασχολούνται με τη στρατηγική το βλέπουν έτσι. Και χρειάζεται αυτή η προσπάθεια να μην έχει μόνο πολιτικό πλαίσιο, αλλά χρειάζεται πολύ βαθιά πολιτισμική ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή. Ευχαριστώ του εμπειρογνώμονε μα, ευχαριστώ του εισηγητέ, ευχαριστώ τον πρόεδρο τη αντιπροσωπείας. Η συνάντηση υπήρξε άκρο ενδιαφέρουσα, αναπτύχθηκαν πολύ σημαντικά θέματα και κρίνει με αιτιολογημένη επιθυμία αναπτύξεως των σχέσεων αυτών και ίσως να μην πετύχουμε στα επόμενα 20 χρόνια πολύ πιο σύντομα να υπογράψουμε αυτή τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. 18 Νοεμβρίου, το λέω για τους συναδέλφους που ίσως ενδιαφέρονται, οι παρόντες, καλέσαμε τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στη Σαουδική Αραβία που καλύπτει και τις σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου για μια ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, προπαρασκευάζοντας τις εκθέσεις των συναδέλφων Μποντής και Νταβίτ. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά όλους. το διάλειμμα για να αλλάξουμε θέση εδώ στα έδρανα και μετά θα ξεκινήσουμε την ακρόαση του Υπουργού της Ουκρανίας. Για τρία λεπτά διακόπτεται η συνεδρίαση. Bene, cari Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων, όπως ξέρετε, με κύριο Κωνσταντίν Κριτσένκο, Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας. Ε, πραγματική χαρά για μένα, κύριε Υπουργέ, ονόματι όλων των συναδέλφων, να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας, όπως γνωρίζετε το κοινοβούλιο μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να αναπτύξει στενότερες σχέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χώρα σας. Παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις πολιτικές εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία και αυτό το βλέπετε διότι εδώ και μερικές εβδομάδες ο κ. Παύλο Κλίμκιν η υφυπουργός σας ε, ήρθε εδώ και ο πρόεδρος Επιτροπής Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Μπόρις Τάρατσουκ, ε, τον συνόδευε. Η παρουσία σας σήμερα μας δίνει μια σημαντική ευκαιρία να μάθουμε από μια άμεση πηγή της προετοιμασίας, ε, προετοιμασίες που κάνει η κυβέρνησή σας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ουκρανίας και θέλουμε να γνωρίσουμε και ποιοι είναι οι στόχοι της κυβερνήσεώς σας. Τι στόχους θέλει να πετύχει η κυβέρνησή σας σε αυτή την σύνοδο. Να προσθέσω και κάτι που μας ενδιαφέρει ως ιδιαίτερος. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας στη χώρα σας θα λάβουν χώρα οι εκλογές, οι δημοτικές δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το γεγονός που αφορά τη διαδρομή της Ουκρανίας προς την ευρωπαϊκή προσχώρηση και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί σας ποιο είναι το πολιτικό κλίμα εντός του οποίου θα διενεργηθούν οι εκλογές. Έχουμε, θα έχουμε και τη χαρά να γνωρίσουμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της κυβερνήσεώς σας. Δυστυχώς έχουμε μόλις μία ώρα για να συνομιλήσουμε μαζί σας, κύριε Υπουργέ, για να δώσουμε και δυνατότητα στους συναδέλφους που σίγουρα θα ενδιαφέρονται πάρα πολύ να σας θέσουν ερωτήσεις και να σχολιάσουν τα όσα θα μας πείτε. Θα σας παρακαλούσα αν έχετε, αν έχετε την καλοσύνη να συγκεντρώσετε την παρέμβασή σας εντός ενός δεκαλέπτου και από τώρα σας παρακαλώ συνάδελφοι, έχει παραπάνω από δύο λεπτά για τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο λακωνικός γίνεται θα σας παρουσιάσω μερικά σημεία που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά για να διαρθρώσουμε την συζήτησή μας. Για την Ουκρανία, η ένταξη με την, προς την Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική προτεραιότητα, όπως φαίνεται, και μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον πρόεδρο Γιαννούκοβιτς. Και στην νομοθεσία μας για εξωτερική πολιτική αναφέρεται ως βασική προτεραιότητά μας η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά για κάτι τέτοιο θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε και σημαντικές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και να συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα, τα κοινωτικά θεσμικά όργανα. Φυσικά, μέχρι στιγμής έχουμε ε, υλοποιήσει πολλά επιτέγματα. Καταρχήν πολιτική σταθερότητα. Με την νέα ηγεσία τέθηκε τέρμα στην αστάθεια και στην θεσμική σύγκρουση χάρη σε μια εδραίωση της εξουσίας. Και εδώ μιλάμε για εδραίωση της εξουσίας, όχι για μονοπόλιο της εξουσίας. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό η υλοποίηση των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων στους χαλεπούς καιρούς που πέρασε η χώρα μας. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς στο διαχωρισμό μεταξύ της, ε, του μονοπωλίου της εξουσίας και της εδραίωσης της εξουσίας. το κοινοβούλιο μας ε, συγκροτήθηκε ε, με βάση το Σύνταγμά μας και με βάση την αρχή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Έχουμε μια αποτελεσματική αλυσίδα εξτελεστική εξουσίας και έχουμε μια σωστή θεσμική διάρθρωση που σέβεται τις δημοκρατικές αρχές, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Η δημόσια διοίκηση έχει αναλάβει πλέον την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία. Σε πέντε μέρες θα λάβουν χώρα οι δημοτικές εκλογές κάτι που θα αποδείξει ότι ζούμε σε μια δραστήρια δημοκρατική κοινωνία. Οι πολίτες μας θα κάνουν τις επιλογές τους όπως σε οποιαδήποτε άλλη δημοκρατική χώρα. Σε πολλές περιπτώσεις η ε, Ουκρανία έχει διατρανώσει τη δέσμευσή της ε, για ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές που θα πληρούν τα, τις διεθνείς προδιαγραφές. Και μάλιστα ο εκλογικός μας νόμος ε, προσαρμόστηκε στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές αποφασίσαμε για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την δημοκρατικότητα των εκλογών μας να προσκαλέσουμε αντιπροσωπείες, διεθνείς αντιπροσωπείες παρατήρησης των εκλογών μας. Επίσης, εφαρμόζουμε συνολικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και μάλιστα τον Οκτώβριο το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε την ε, μεταρρύθμιση του 2004 και επανέφερε το νομικό πλαίσιο του συντάγματος του 1996 που πρόβλεπε ε, την Ουκρανία ως προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Υπάρχει συνένεση στην Ουκρανία ότι οι συνταγματικές αλλαγές του 2004 ε, παραβίαζαν τις θεσμικές διαδικασίες αποφεύγοντας οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση και παραβίαζαν το κράτος δικαίου. Αυτό ήταν η γνώμη και πολλών Ουκρανών πολιτικών. Και εξυπηρετούσε αυτό το εσφαίρετο του ε, αρχηγού της αντιπολίτευσης και του βασικού κόμματος αντιπολίτευσης. Τώρα με τους 30 νέους νόμους ε, που υιοθετήσαμε ε, υλοποιούμε την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου και προσπαθούμε να γεφυρώσουμε όλα τα κενά που υπήρχαν στην νομοθεσία. Βέβαια δεν σταματούν εδώ τα πράγματα και οι προσπάθειές μας. Θα συνεχίσουμε με την βελτίωση του συστήματος των εξουσιών. Δηλαδή θα ακολουθήσουν και νέες αλλαγές που θα γίνουν με επαγγελματικό, ανοιχτό τρόπο, χωρίς να περιθωριούμε κανένα με την τρίτη εδραίωση του κράτους δικαίου, τη δικαστική μεταρρύθμιση και την πάταξη της διαφθοράς, θα υλοποιήσουμε τις βασικές προτεραιότητες της Ουκρανίας. Παρά κάποιες αποφάσεις που χαρακτηρίστηκαν επίμαχες, σημειώνουμε πρόοδο στους προηγούμενους τομείς. Και μάλιστα η πρόσφατη έγκριση νομοθεσίας για το δικαστικό κλάδο θα εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας σε συνεργασία με την ε, Επιτροπή της Βενετίας με στόχο να υλοποιήσουμε υψηλές προδιαγραφές ε, για την ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης, πρόσβαση στη δικαιοσύνη όλων των Ουκρανών πολιτών, των κατοίκων της Ουκρανίας και την πάταξη της διαφθοράς. Επίσης, θέλουμε να βαθμίσουμε τα μέσα και τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της θωροδοκίας. καταφέραμε να αναχαιτήσουμε την οικονομική κατά βαράθρωση της Ουκρανίας και μάλιστα για το πρώτο εξάμεινο του χρόνου η αύξηση του έπειτα ήταν 6% και η μηχανική παραγωγή σημείωσε μια αύξηση του 12%. Και μάλιστα ε, εφαρμόσαμε πολλές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα η οθεσία της νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες, πιστοποίηση και μάλιστα κύρωση πολλών διεθνών ε, συνθήκων για τη μετανάστευση συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και προσπάθεια διεκπαιρέωσης των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Όλες αυτές είναι σημαντικές για να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, οι μεταρρυθμίσεις αυτές ε, χαράζονται και εφαρμόζονται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να προχωρήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση με την στενή συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα με ιδιαίτερη χαρά να σας ενημερώσω για, για την πρόοδο της Ουκρανίας ό,τι αφορά τα βασικά έγγραφα για τις μεταρρυθμίσεις που είναι κλειδί για τις μεταρρυθμίσεις της Ουκρανίας και μέχρι στιγμής έχουμε εφαρμόσει 10 από, τις 15, 10 από τα 15 μέσο και πρόθεσμα ε, μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το Matrix, το βασικό όργανο. Επίσης, βελτιώνουμε και το επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας. Προσπαθούμε να επιλύσουμε το μακροχρόνιο πρόβλημα της επιστροφής του ΦΠΑ. Επίσης προσπαθούμε να βελτιώσουμε, να απλοποιήσουμε το φορολογικό σύστημα, να μειώσουμε τη φορολογική πίεση και να εφαρμόσουμε τις συστάσεις των Ευρωπαίων εταίρων μας για τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα. Βέβαια, χρειαζόμαστε στην Ουκρανία ακόμη πολλή προσπάθεια και πολύ δρόμο να διανύσουμε. Το θέμα της ε, ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας στο μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου εκπρόσωποι του ΕΣΕ για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης πραγματοποίησαν ε, επίσκεψη στην Ουκρανία για να δημιουργήσουν μια ε, εξέταση της κατάστασης στην Ουκρανία εκφράστηκε η ε, αναγνώριση της προσπάθειας της Ουκρανίας για την εξασφάλιση της ε, ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν και ασκήθηκαν και κάποιες επικρίσεις που φυσικά θα τις λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Οι Ουκρανικές αρχές είναι έτοιμες ε, να λάβουν υπόψη και να εφαρμόσουν και τις συστάσεις της κοινοβουλευτικής τη κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη ε, με βάση το ψήφισμα 1755 του Οκτωβρίου του 2010. Φυσικά θέλουμε να ελοπίσουμε το κράτο δικαίου, τη δημοκρατία και το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι κοινέ αξίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και που είναι κλειδί για την εμβάθυνση των σχέσεών μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω, η, ένταξη, η εμβάθυνση της, ε, των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Ουκρανική ηγεσία. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια και για το πρόγραμμα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανική ηγεσία πιστεύει ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση σημαίνει καταρχήν εφαρμογή των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία με βάση τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το βασικό καθήκον ε, των διαφόρων επιπέδων εξουσίας είναι να οριστικοποιήσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις για τι συμφωνίε σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την υλοποίηση του, της ζώνης ελευθέρου εμπορίου με αμοιβαίω επωφέλη βάση και με ένα λογικό χρονοδιάγραμμα. Και οι δύο συμβαλόμενε πλευρές καλούνται να, υλοποιήσουν, να οριστικοποιήσουν, διεκπαιρέσουν διαπραγματεύσει ό,τι αφορά την Συμφωνία Σύνδεσης. επειδή έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτό το πολιτικό σκέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας μένει το οικονομικό σκέλος της Συμφωνίας Ελευθέρω Εμπόριου, FTA. Επίσης θέλουμε να εμβαθύνουμε τις οικονομικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμής ήταν στόχος μας η συνεργασία, αλλά τώρα είναι περισσότερο στόχος μας η ένταξη και θέλουμε ένα είδος πολιτικής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οικονομικής ολοκλήρωσης. Θέλουμε εμβάθυνση των θεμάτων στα πράγματα του DCFTA. Θέλουμε επίσης να κρατήσουμε υψηλό το επίπεδο των φιλοδοξιών μας ό,τι αφορά την μελλοντική ζώνη ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να είναι όσο πιο φιλόδοξη γίνεται, γιατί είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Γιατί έτσι θα έρθει και η Ουκρανία πιο κοντά από οικονομική άποψη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να επίσης την προσοχή σας και σε ένα άλλο ε, θέμα, το θέμα της απελευθέρωσης ε, των ε, θεωρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για τους Ουκρανούς πολίτες και για την Ουκρανική ηγεσία. Συμφωνούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι κατά παράδοξο τρόπο 20 χρόνια μετά την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου δεν έχουμε ακόμη αποκαταστήσει τις την κατάσταση ό,τι αφορά τις ε, θεωρήσεις. Ε, υπάρχει ακόμη το τείχος των θεωρήσεων. Δεν μπορούν οι Ουκρανοί πολίτες να ταξιδεύουν ελεύθερα από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία απελευθέρωση αυτού του καθεστώτος, ε, καθεστώτος θα είναι απτή απόδειξη της αίσιας έκβασης των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρυσι με τη σχετική νομοθεσία για τη συνεργασία δικαιοσύνης και εσωτερικών ε, κάναμε ένα βήμα προς την κατάθεση των μεταρρυθμίσεων και σας ευχαριστούμε για τη χθεσινή, μας, για τη σας απόφαση που σημείωσε πρόοδο στο θέμα αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της σημερινής συζήτησης αξιότιμη Ευρωβουλευτέ θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ την ε, αρχική μου παρουσίαση και να σας πω ότι περιμένω με ανυπομονησία τις ερωτήσεις σας και την περαιτέρω συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κόβολ, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο κ. Χόβαλ, Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ουκρανίας. Για δύο λεπτά παρακαλώ, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι η προηγούμενη εβδομάδα ήταν από τις πιο πολυτάραχες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν συζητήσαμε το ψήφισμα και για την Ουκρανία. Χαίρομαι που η, η Ουκρανική διπλωματία τις τελευταίες εβδομάδες είναι πολύ δραστήρια και ενεργή και ελπίζω ότι με τις πολιτικές αυτές αλλαγές και τις επερχόμενες εκλογές θα φτάσουμε σε ένα σημείο καμπής και θα βελτιωθεί και η εντύπωση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία. Είχαμε, θα, έχουμε και την ε, αποστολή παρατήρηση των ε, εκλογών, αλλά και την επόμενη, συνεδρίαση επόμενης εβδομάδας. Θα ήθελα να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις. Με ποιον τρόπο, από θεσμική άποψη, συντονίζει η Ουκρανική κυβέρνηση τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κάποια ειδική επιτροπή, υπάρχει κάποιο ειδικό σώμα. Πώς ε, βλέπετε τον, καλύτερο θεσμικό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ Προέδρου και Κυβέρνησης. Κατά τη γνώμη σας, ε, πώς μπορείτε να συσπηρώσετε όλες τις πολιτικές δυνάμεις υπέρ της ε, προοπτικής της ένταξης. Ξέρουμε και από την εμπειρία της, πολι... της Πολωνίας και άλλων ανατολικών χωρών ότι υπήρχε ένα πολιτικό σώμα που προσπαθούσε να συντονίσει όλες τις πολιτικές ε, δυνάμεις προς το στόχο της... Ε, των σχέσεων και της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι μετά τις εκλογές και την συνάντηση που θα έχουμε στο Κίεβο θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να συγκροτηθεί ένα τέτοιο σώμα. Και νομίζω θα είναι συνέχεια και τη συζήτηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Χόβαλ. Ο κύριος Μπρόκ έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Πρόεδρε, ο... ευχαριστώ τον Υπουργό που βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα και έχω τρία σύντομα ερωτήματα. Πιστεύετε ότι υπάρχει ευκαιρία η ανατολική εταιρική σχέση να διαμορφωθεί με πολυ... πολυ Να υπάρξει δηλαδή συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο και όχι μόνο με κάθε χώρα ξεχωριστά. Κατά δεύτερον, πώς θεωρείτε... Ποιες προτάσεις έχει να κάνει προς την κατεύθυνση αυτή η Ουκρανία, γιατί θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι και το ΕΛΚ πέρα από τις επικριτικές ε, διαθέσεις σε πολλές περιπτώσεις ε, θεωρεί ότι η θέση της Ουκρανίας είναι στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις θεωρήσεις το TGZFTA μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου δηλαδή μια μορφή και αυτό προκειμένου για αποτελέσματα με γρήγορο τρόπο γιατί ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε μόνο Ένωση Οικονομική, αλλά και Ένωση Αξιών. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι υπάρχει ε, σταθερότητα στην Ουκρανία, πολιτική σταθερότητα, με σαφές ε, εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά αυτή η σταθερότητα ε, επιτυχάνεται μόνο με εκ των έσω, όχι με ρυθμίσεις. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει την ημέρα των εκλογών, αν για παράδειγμα όμως ε, δεν μπορεί κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να εκφραστεί. Αυτό δεν κινείται προς την σωστή κατεύθυνση της εμπιστοσύνης. Ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν δικαστήρια για να εκδοθούν αποφάσεις που θα καθιερώσουν την πλειοψηφία. Δεν είναι στόχος ε, για μένα να ε, επαναγκαθιδρυθεί το Σύνταγμα του 96. Θα πρέπει να διασφαλίζουμε καταρχάς την εξαρτησία των αρχών αυτών. Σας ευχαριστώ κύριε Μπροκ. Για δύο λεπτά ο κύριος Σίβιετς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. τελείως τυχαία είχα σκεφτεί και εγώ τα ίδια που είπε ο κύριος Μπροκ και αυτό θα συνεχίσω κατά κάποιο τρόπο τη σχέση του. Θα πρέπει να βγούμε αυτό το θεσμικό αδιέξοδο, γιατί η συζήτηση για το Σύνταγμα της Ουκρανίας είναι ένα σύριαλ. Ένα σύριαλ το οποίο είδαμε την αρχή αλλά δεν βλέπουμε το τέλος. Πάντα το Σύνταγμα είναι το μήλο της έριδας και όποιος έχει την εξουσία θέλει να αξιοποιήσει το Σύνταγμα για το συμφέρον του. Φυσικά αυτό δεν συμβαίνει, αλλάζει το πολιτικό κλίμα και δημιουργείται μία μόνιμη σύγκρουση. Ήταν και πολωνική αυτή η εμπειρία, αλλά τελικά είναι οικουμενικό φαινόμενο. Χρειάζεται να αναλυθεί μία πρωτοβουλία από την πλειοψηφία, από την κυβέρνηση και τον πρόεδρο Χαίρομαι για την εδραίωση της εξουσίας, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα αυτή την εδραίωση της εξουσίας, αλλά αν είναι γεγονός αυτή η εδραίωση, τότε με ποιο τρόπο θέλετε να ξεπεράσετε αυτό το αδιέξοδο της, του συντάγματος, αν αποκλείσετε την αντιπολίτευση από τη συζήτηση. Είναι αδύνατο να επιληθεί το συνταγματικό διέξοδο αν δεν συμπεριλάβατε και την αντιπολίτευση στις διαπραγματεύσεις για το Σύνταγμα και στις συζητήσεις. μερικές φορές αναφέρονται κάποια νομικίστικα επιχειρήματα, αλλά αυτό είναι σαν φαρσοκομωδία. Γιατί για πολλά χρόνια ε, χώρα ε, έμενε, ε, στηριζόταν σε ένα ιονί σύνταγμα, όπως φάνηκε και από την ακύρωσή του. Νομίζω ότι για να εξασφαλιστεί μια σταθερότητα και μια μονιμότητα της εξουσίας, χρειάζεται μια εδραίωση και μια επίλυση του στεγματικού αδιεξόδου στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βιέτς. Νέιτς. Θα θα πάρει το λόγο. Κυρία Νέιτς, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε λοιπόν. Εξωτερική πολιτική αφορά το ερώτημά μου. Η εικόνα που παρουσιάζεται πολύ συχνά είναι ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα δίλημα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ρωσία. Είτε το ένα είτε το άλλο. Είτε θα υπάρξει προσέγγιση προς τη Ρουσία, άρα αποστασιοποιείται την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ανάποδο. Πείτε μας πώς το βλέπετε εσείς το θέμα. Sí. Σας ευχαριστώ κυρία Νέιτς. Κύριος Γκάλερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Η χώρα σας ε, πρέπει να ανταπεξελθεί στις ε, προκλήσεις για να εξασφαλίσει η καλή ζωή στις πολίτες της. Εμείς σας ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σας ε, υποστηρίζουμε. Και συχνά έχουν ακουστεί ανησυχίε μας ωστόσο στο Κίεβο, αλλά το ψήφισμα της 5ης Οκτωβρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχει επιπτώσεις ε, στη χώρα σας. Ποια μέτρα θα ληφθούν, ποια ε, μέτρα έχουν ληφθεί για να καταστεί δυνατή και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του κόμματος κ. Τιμοσέγκο στις εκλογές. Μιλάμε για ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν και αμφισβητώ κατά πόσο οι εκλογές οι δημοτικές μπορούν να θεωρηθούν ελεύθερες και δίκαιες. Ε, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Ρουμανία που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύουν ότι ο δρόμος για την εξασφάλιση του πολίτη δεν περνάει μέσω των ολιγαρχιών και του αυταχειρισμού, αλλά μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της δημοκρατίας. Ελπίζω και το Σοσιαλιστικό Κόμμα στο σημείο αυτό να ε, χρησιμοποιήσει την εξουσία της προς αυτήν την κατεύθυνση. Μία ερώτηση Είχα πει προηγουμένως ε, στην ε, γραμματεία να χρησιμοποιήσει το ουκρανικό αλφάβητο για το όνομά σας μπροστά εδώ. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εσείς ποια ε, γλώσσα προτιμάτε. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Κύριος Χάρμς για δύο λεπτά. Η κυρία Άρμς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να εκφράσω ότι με την απόφαση να μην ψηφίσουμε το ψήφισμα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι έχουν διεκπεραιωθεί τα σημεία τα επικριτικά που συμπεριλαμβάνονται στο ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρα από το φάσμα των πολιτικών ομάδων που συνδέονται ενδεχομένω με τα κόμματα στην ε, Ουκρανία προσπαθεί να διαμορφώσει μια εικόνα για το τι γίνεται στην περιοχή και ποιε ανησυχίες είναι δικαιολογημένε. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω, γιατί το έθεσε το ερώτημα και ο κύριος Γκάλερ, να μας εξηγήσετε γιατί ο εκλογικός νόμος ε, χρειάστηκε να αλλάξει πριν από τι δημοτικέ εκλογέ και γιατί θεωρήθηκε σωστό στην περιοχή να διαμορφωθεί ο νόμος αυτός με τέτοιο τρόπο προκειμένου πολλές τοπικές οργανώσεις και μη κυβερνητικέ οργανώσεις σήμερα να μην έχουν τη δυνατότητα να κατέβουν υποψήφιες για τις εκλογές αυτές. Αυτό είναι σημαντικό το ερώτημα και σε ό,τι αφορά την δημοκρατική εξέλιξη, δημοκρατική πρόοδο σε τοπικό επίπεδο. Πέραν αυτών, μας απασχόλησε ιδιαίτερα ο νέος ρόλος των μυστικών υπηρεσιών στην Ουκρανία. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε, εσείς ο ίδιος, πώς αντιδράτε στις κατηγορίες αυτές. Ο νέος αυτός ε, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών ασκεί όλο και πιο μεγάλη πίεση στα μέσα και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Ουκρανία και όχι μάλιστα μόνο στην Ουκρανία αλλά και σε οργανώσεις όπως ε, το Ίδρυμα Κόνοντα Αντενάουερ ή Ζόρος που δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Ουκρανία. Εκτός αυτών μας ε, αναφέρθηκε ότι οι μυστικοί υπηρεσίε στην Ουκρανία έχουν αναλάβει δράσεις κατά τεσσάρων ε, δημοσιογράφων. Δεν πρόκειται να τους αναφέρω ονομαστικά. Ο κ. Κλιμέντια, είναι ένας από αυτούς. Πείτε μας λοιπόν την ε, αντίδρασή σας για τις κατηγορίες αυτές και κάτι άλλο που μας απασχολεί. Υπάρχει ένα κύμα συλλήψεων των πρώην ε, μελών της κυβέρνησης Τιμοσέγκο και αυτό είναι ένα σήμα, μια ένδειξη ότι εξακολουθεί να μένεται μια πολύ αντιφατική κατάσταση στην ε, Ουκρανία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κυρία Χάνς. Πέτερινγκ είναι το επόμενο όνομα που έχω μπροστά μου. Για δύο λεπτά και ως Πέτερινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών. Να σας ρωτήσω το εξής. Πριν από δύο χρόνια ως πρώην πρόεδρος της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχα την ευκαιρία να εκφράσω τη θετική μου άποψη για την Ουκρανία στο δικό σας κοινοβούλιο, αλλά σήμερα ε, είναι πολλές οι ανησυχίες που επικρατούν και συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Σημειώσαμε την ε, υπόθεση ενός δημοσιογράφου κατά πάσα πιθανότητα του ιδίου που ανέφερε και η συνάδελφος Χάρμς. Ο δημοσιογράφος αυτός λοιπόν του αφαιρέθηκε ο υπολογιστής του και όπως μας ανέφεραν ε, τα ανακοινοθέντα, στον υπολογιστή αυτόν είχε και το διδακτορικό του. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Και εμείς ε, έχουμε την εντύπωση ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς ε, περιορίζεται ή μάλλον ε, εστιάζεται στους κόλπους της αντιπολίτευση. Θα ήσασταν πολύ πιο αξιόπιστοι ότι θα αν εξετάζονται και θέματα που πλήττουν την ίδια την κυβέρνηση. Και τέλος, θα ήθελα να αναφέρω το εξή χωρί να εμβαθύνω, Μια και η συνάδελφο ανέφερε το Ίδρυμα Κόνραντ Άντεναουερ, ότι θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις σχετικές με ιδιαίτερη ανησυχία. Θέλουμε συνεργασία με την Ουκρανία, αλλά με τη βάση μιας ε, εξέλιξης κράτους δικαίου. Σας ευχαριστώ κύριε Πέτερινγκ. Για δύο λεπτά κύριε Σεβερίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, είσαστε υπουργό Εξωτερικών και πολλές από τις ερωτήσεις μας αφορούν θέματα εσωτερικών. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα και εγώ να πω, πριν σας θέσω ένα ερώτημα, ότι έχουμε αναβάλει την απόφασή μας επί του ψηφίσματος για την Ουκρανία, όχι γιατί θέλουμε να εθελοτυφλούμε όσον αφορά τις ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν στην Ουκρανία, αλλά επειδή θέλουμε να ανοίξουμε ακόμα πιο ανοιχτά τα μάτια μας όταν πρόκειται να λάβουμε απόφαση και θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες για να ξέρουμε ακριβώ ποιες είναι οι διαδικασίες, τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορούμε να πούμε περί όλων αυτών. Ταυτόχρονα, επανερχόμενος στις ερωτήσεις, νομίζω ότι η διπλωματία είναι η δυνατότητα να συντεριάζει τα αντίθετα καμιά φορά. Λοιπόν, ερώτηση. Επιχειρηματικά συμφέροντα και πολιτικές δομές πώς μπορείτε να ταιριάξετε στη χώρα σας ή μάλλον πώς θα μπορούσατε να, διαχειρι... διαχωρίσετε τη διαμόρφωση πολιτικής από τις επιχειρήσεις. Δεύτερη ερώτηση. Πώς βλέπετε τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα σας όσον αφορά την αποκέντρωση. Επίσης, πώς βλέπετε τις μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών. Η κυβέρνησή σας μπορεί να συνεργαστεί με όλες τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου μας ανεξαρτήτως πολιτικών προσανατολισμών. Μπορείτε να εξισορροπήσετε τις ανατολικές και δυτικές εξωτερικές σας σχέσεις, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι υπέρ της Ουκρανίας και υπέρ της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και της Συνεργασίας επίσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ρωσίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σεβερίν. Για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Λίζα. Ε, Σας ευχαριστώ. Με διευκολύνετε κάπως κύριε Υπουργέ και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα και το επίμαχο ζήτημα της επιστροφής του ΦΠΑ για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και τις πολωνικές κυρίως που εξάγουν. Αλλά όπως είπατε βρίσκεται σε σωστό δρόμο διευθέτηση το ζήτημα της επιστροφής του ΦΠΑ. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω και κάτι για την εξωτερική πολιτική, γιατί υπουργός εξωτερικών είστε. Οι Ουκρανικές αρχές ε, υποστήριξαν και το όραμα άλλο, ε, στερνίζονται και άλλα οράματα, ε, υποστηρίζουν και άλλες χώρες για τα όραμά τους της Ευρωπαϊκής Ένταξης και της ένταξης στο ΝΑΤΟ, όπως της Γεωργίας. Σε ό,τι αφορά αυτή την ευρωατλαντική προσδοκία άλλων χωρών, μεταξύ άλλων και της Γεωργίας, ποια είναι η δική σας θέση. Επίσης, ποια είναι η θέση της κυβέρνησής σας σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Λευκορωσία, εν ώψη των ε, περχόμενων εκλογών που θα λάβουν χώρα στη Λευκορωσία. Εμείς έχουμε πολλές επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την τήρηση των δημοκρατικών αρχών για τις ε, λευκορωσικές εκλογές. Ευχαριστώ κύριε Λίσεκ. Μίσκι είναι το επόμενο όνομα. Κύριος Μίσκι, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Γκρισέγκο. Από ό,τι γνωρίζω, ο Στέφαν Μπαντέρα ανακηρύθηκε ήρωα, ήρωας της Ουκρανίας. Συμμετείχε στο ολοκαύτωμα από ό,τι γνωρίζω. Ήταν αντισημιτικό, αντισημίτης όσον αφορά την προσέγγιση του και αυτά που έλεγε. Ποια είναι η απόψή σας, είναι ήρωας ή εγκληματίας. Και τι σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνησή σας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Μίρσκι. Ο κύριος Λαντσμπέργκης έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Κύριε Υπουργέ, στη χώρα σας τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται προσπάθειες, προσπάθειες για να ενισχυθεί η Ουκρανική γλώσσα στην δημόσια ζωή και στην εκπαίδευση. Και αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο κατά την Προεδρία του κ. Γιουσένκο. Και πολλοί κατηγορούν την Ουκρανία για το γεγονός αυτό. Υπό την κυβέρνηση του κ. Γιαννουκοβίτς ε, γίνονται κατηγορίες, ακούγονται κατηγορίες για την ε, εκδίωξη της γλώσσας, ότι χάνεται δηλαδή ο κρονικός χαρακτήρας. Σχολιάστε παρακαλώ. Αληθεύουν αυτές οι κατηγορίες και πρόκειται για μια διάθεση σεμιβασμού, αν θέλετε, και επαναχώρησης έναντι της Ρωσίας. Υπάρχει μια τέτοια τάση εκδίωξης του κρανικού στοιχείου ή μήπω είναι απλά αιτιάσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Λαντμπέργκης. Ο κύριος Σούλτς κλείνει το γύρο των ερωτήσεων για δύο λεπτά. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε στην αρχή για τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προοπτική. Να σας θέσω ένα ερώτημα ο πλευράς πολιτικής ασφάλειας με την παράταση της, της παραμονής του ρωσικού στόλου στην Κρυμαία. Θεωρείτε ότι ο κίνδυνος Υπάρχει κάποιο κίνδυνο και ποιε είναι οι σχέσει, ποια είναι η αντιμετώπιση σα ε, το, στο ΝΑΤΟ για την πιο έντονη αυτή στρατιωτική σχέση, η οποία φτάνει μέχρι τα μέσα του αιώνα. Ποιε είναι οι προπτικέ που έχετε με το ρωσικό στόλο. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε το βάρος το να απαντήσετε σε 11 παρεμβάσεις σε λιγότερο από 10 λεπτά. Βέβαια μπορείτε να έχετε κάνα δύο λεπτά και παραπάνω, αλλά σας παρακαλώ αν, είστε, αν είναι δυνατόν να είστε σύντομος. ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που θα ήθελα να αναπτύξω τις απαντήσεις αυτές ερωτήσεις. Αλλά έχοντας συνηθίσει να απαντώ λακωνικά, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Να ξεκινήσω με το τι γίνεται στην Ουκρανία όσον αφορά τις εκλογές και να απαντήσω σχετικές ερωτήσεις. Και επίσης όσον αφορά το θέμα το συνταγματικό στη χώρα. Πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε πολλές δηλώσεις στις οποίες αναφέρεται στην ανάγκη διεξαγωγής δικαίων εκλογών που θα συμμορφώνονται με τις υψηλότερες ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Γι' αυτό καλέσαμε όλους αυτούς τους παρατηρητές από διάφορες ε, διεθνείς μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ο πρόεδρος μου συναντήθηκε μόλις πριν από μερικές ώρες και είναι ένας τρόπος αυτός με τον οποίο στέλνουμε μήνυμα προς τους φίλους μας στον κόσμο και στην Ευρώπη πόσο σοβαρή μας αφορά τη διεξαγωγή ανοιχτών και δικαίων εκλογών. Μια δημοκρατία σε, μετάβαση είναι μια πρόκληση και αποστολή. Και είναι μια αποστολή που έχει πάρει πολύ στα σοβαρά και η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος. Και γι' αυτό μετά από την αρχική παρουσίαση του νόμου για την τοπική αυτοδίκηση, μάλλον την ψήφιση του νόμου για την τοπική αυτοδίκηση, τις τοπικές εκλογές, έγιναν και αλλαγές που αντικατοπτρίσαν τις επικρίσεις που είχαν ακουστεί και επετράπηκε η συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων. Αλλάξαμε τον νόμο γιατί ο παλιό ήταν άδικος. Ακούμε τις επικρίσεις, υπάρχει διάδραση, διαδραστική σχέση και με την αντιπολίτευση και με την κοινωνία των ε, πολιτών στην Ουκρανία. Δεν επιβάλλουμε τις απόψεις μας, αλλά προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη τη γνώμη της πλειοψηφίας εκείνων που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία και του ίδιου του λαού βέβαια. Θα ήθελα να πω ένα-δύο λόγια για το Σύνταγμα. Όταν επιστρέψαμε, επιστρέψαμε στο Σύνταγμα το 1996, δεν έγινε αυτό διότι το αποφάσισε η κυβέρνηση αλλά διότι 18 από τα 18 μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, 17 ε, ψήφισαν υπέρ της επιστροφής και στο παλιό Σύνταγμα και της ανάκλησης αποφάσεως των αποφάσεων που ελήφθησαν το 2004 που είχαν παραβιάσει και τους συνταγματικές ε, διατάξεις και το νόμο γενικότερα. Και ήταν ο μόνο φορέ που πάρει αυτή την απόφαση το Συνταγματικό Δικαστήριο, όχι η κυβέρνηση. Και εγώ, σαν μέλο τη κυβερνήσεω, δεν μπορώ να συζητήσω την απόφαση του φορέα αυτού. Είχαμε μόνο μία επιλογή να εφαρμόσουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Και έτσι πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος σε κάθε δημοκρατική χώρα. Θα ήθελα εδώ να σας παραθέσω κάτι, να σας αφέρω κάτι από τα πορίσματα της Επιτροπής της Βενετίας για το Σύνταγμα της Ουκρανίας, μελέτη που έγινε το 1996. Το Σύνταγμα λέει δημιουργεί ισχυρή εκτελεστική εξουσία και έχει σύστημα ελέγχων ούτω ώστε η επιστροφή σε αυταρχικό καθεστώς είναι κάτι αδύνατον. Το κράτος δικαίου υποστηρίζεται από το Σύνταγμα υποστηρίζεται τοπική αυτοδιοίκηση και δίνεται ε, σημαντικός ρόλος συνταγματικό δικαστήριο και δημιουργεί έτσι μια, ένα δημοκρατικό πολιτισμό, μια δημοκρατική νοοτροπία στην Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, σημαντικές απόψεις αυτές, σημαντικό το πόρασμα από τον πιο έγκυρο φορέα στον τομέα. Αλλά όπως προανέφερα στην αρχική μου παρουσίαση, δεν έχουμε σταματήσει εδώ. Πιστεύουμε ότι περαιτέρω βελτιώσεις πρέπει να γίνουν αλλά θα αποφασιστούν μέσω μιας διαδικασίας στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, θα μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους. Έχουμε σημαντικό πρόβλημα στη χώρα μας ότι δεν μπορεί μία μόνο πολιτική δύναμη να συμμετέχει. Αλλά συμφωνώ ότι κάποτε στην Ανατολική Ευρώπη οι πολιτικές δυνάμεις στις περισσότερες χώρες ενώθηκαν γύρω από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δυστυχώς, εμείς βλέπουμε πολιτική κίνηση προς την Ευρώπη μόνο όταν ηγείται αυτή η πολιτική δύναμη. Όταν δεν ηγείται αυτή η πολιτική δύναμη, όλα γίνονται για να σταματήσει η διαδικασία. Τίθεται εμπόδια. Αυτό συμβαίνει, διότι δεν υπάρχει παραγωγικός διάλογος στην χώρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι καμιά, να το συζητήσουμε εκτός χώρας. Γι' αυτό ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσεφέρθη να συναντηθεί με τον κύριο Μάρτιν στι 30 ε, Οκτωβρίου, δεν υπήρξε απάντηση. Πώ μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση αν δεν να συναντηθεί με εκείνου που στέλνουν μηνύματα επί διαφόρων πτυχών που αφορούν τη ζωή στην Ουκρανία, εγώ ήμουν έτοιμο να συνομιλήσω σήμερα. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις συζητήσει. όταν οι εταίροι μας θα είναι έτοιμοι ανεξάρτητα από το πολιτικό, πολιτική τους κατεύθυνση. Δεν κάνουμε επιλογή πολιτικών κομμάτων. Πιστεύουμε ότι όλοι όσοι κάθονται εδώ είναι φίλοι μας, είναι εταίροι μας έχουν ανησυχίες νόμιμες καμιά φορά, δίκες που πρέπει να καλύψουμε. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να επισκεφθείτε και εσείς την Ουκρανία και ίσως να έχετε χρόνο να συναντηθείτε και εσείς με όλους τους εκπροσώπους της Ουκρανίας και από την αντιπολίτευση και από την ε, κυβέρνηση. Δεν εκπροσωπώ καμία πολιτική δύναμη, εκπροσωπώ την κυβέρνησή μου υπό την ιδιότητά μου ως υπουργό και θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια θέματα που αφορούσαν τις αποφάσεις που ελήφθησαν εδώ. Η καθυστέρηση του ψηφίσματος για την Ουκρανία ήταν η σωστή απόφαση. Εμείς νομίζω ότι έχουμε δώσει απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που είχαν τεθεί στο Συμβούλιο. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται ε, μια επαφή πριν κρίνει κανείς. Χρειάζεται συζήτηση, ενδελεχής γνώση και πρέπει κανείς να ακούει διάφορες πηγές και διάφορες φωνές. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ενδιαφερόμαστε για μια τέτοια συζήτηση που αντικατοπτρίζει η ευρωπαϊκή παράδοση, την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική παράδοση πιστεύω και είναι και δική μας παράδοση αυτή. Δύσκολα θέματα, όπως αναφέρθηκε, αναφερθήκατε στην επίσκεψη εκπροσώπου του Καθολικού Πανεπιστημίου που έθεσε κάποια ζητήματα που είχαν τεθεί στον Πρίτανη. Τέλο πάντων, τελικά ζήτησε συγγνώμη για αυτά που υπόθηκαν. Έγινε, η κυβέρνηση παίρνει σοβαρά, στα σοβαρά αυτά τα θέματα. Είμαστε σε μεταβατική φάση. Και τα θέματα των επαφών των κυβερνητικών υπηρεσιών και των κυβερνητικών υπαλλήλων ε, τα εξετάζονται. Χρειάζεται αναβάθμιση για να συμμορφωθούμε με τις προδιαγραφές των διαφόρων δημοκρατικών κρατών. Κάνουμε προσπάθειες. Απέχουμε από το ιδεώδες, σας ακούμε και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και να αντιδράσουμε σε σχετικές δικές σας προτάσεις. Όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εμείς ως εκπρόσωποι είτε του Κοινοβουλίου είτε της κυβερνήσεως Όλοι μας θέλουμε, τι θέλουμε να κάνουμε κατά πολέμηση, διαφθορά ή να αφήσουμε κάποιους εκτός. Πιστεύουμε ότι οι πρώην εκπρόσωποι της uh, κυβερνήσεως έχουν ασυλία από έρευνες ή όχι. Να σας πω, οι πρώτες συλλήψεις και οι πρώτες έρευνες δεν είχαν σαν στόχο τα μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης. Η πρώτη σύλληψη έγινε όταν υφυπουργό Οικολογίας συνελήφθη για δωροδοκία. Μετά από λίγες εβδομάδες μόλις, ε, από τότε που διέπραξε κάποιο αδίκημα και μετά από δύο εβδομάδες το αφεντικό του, ο υπουργό που υποστήριξε αυτό τον υφυπουργό, καταψηφίστηκε από την κυβέρνηση, έχασε τη θέση του την κυβέρνηση από τη συμμαχία. Και αυτό συνεχίζεται. Η εκαθάριση των πολιτικών τάξεων δεν έχει σχέση με το πολιτικό χρώμα. Θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Η διαφθορά δεν θα επιτραπεί πουθενά, ούτε και στο δικαστικό κλάδο. Διότι στο δικαστικό τομέα είχαμε μεγάλη διαφθορά, ήταν πηγή αστάθειας και ήταν ανίκανος ο δικαστικός τομέας να υπερασπιστεί τα δίκαια, τα δικαιώματα των πολιτών. Γι' αυτό Ψηφίσαμε αυτό το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Προβλέπει αυτονομία αλλά και ευθύνη των δικαστών. Είναι υπεύθυνοι να καταλήγουν σε αποφάσεις τεκμηριωμένες, δικαιολογημένες βάσει του νόμου. Να μην υπάρχουν άλλα κίνητρα στον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Τώρα, σχέση με τη Ρωσία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να πω κανένα δύο λόγια για αυτό το θέμα διότι ετέθη αυτό το ζήτημα σε μία δύο ερωτήσεις τουλάχιστον. Ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας δεν δημιουργεί καμία απειλή σε κανέναν. Τα περισσότερα σκάφη έχουν ηλικία πάνω από 40 χρόνια και υποτίθεται ότι θα αντικατασταθούν. Είναι πολύ περιορισμένη η δύναμη, δεν είναι απειλή για τον Ατο. Είναι τοπικός στόλος για τοπικές ανάγκες επιστρέφοντας στην εξομάλυνση των συσσωμαλής σχέσεις με την ε, Ρωσία θα υπάρξει και προβλεψιμότητα ε, της πολιτικής εικόνας που θα επικρατήσει στην Ευρώπη. Και έτσι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, όπως και οι σχέσεις Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπουν σε ένα μονοπάτι που θα είναι υποφελές για όλους και θα πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό και είμαι πεπισμένος ότι η Ουκρανία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, συνέβαλε σε αυτή την ε, πορεία. Τώρα, το θέμα των γλωσσών, να απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα. Η Ουκρανική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα στην Ουκρανία. Ε, είναι η γλώσσα του κράτους και θα συνεχίσει αυτό. Υπάρχουν διάφορες απόψεις από διάφορα πολιτικά κόμματα σχετικά με την ισορροπία που θα έπρεπε να επικρατεί. Τι προβλέπει η χάρτα για τις περιφερειακές γλώσσες που υπέγραψαν πάρα πολλές χώρες και ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της γλώσσας του κράτους. Είναι μια συνεχιζόμενη συζήτηση αυτή. συζητείται εκτενώς το θέμα. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Κοινοβούλιο, όχι από την κυβέρνηση. Συνεχίζεται η συζήτηση. Και χρειάζεται ισορροπία. Ισορροπία που θα αντικατοπτρίζει τις ευρωπαϊκές αξίες όσον αφορά το συγκεκριμένο αυτό τομέα. Δεν ξέρω αν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου ή όχι. Θα ήθελα απλώς να πω ένα-δύο πράγματα για κάποιες λεπτομέρειες για την εξαφάνιση δημοσιογράφου του Ντεμέντεφ. Το παίρνουμε πολύ σοβαρά το θέμα. Είναι συμπολίτη μας. Εάν έχει χαθεί η ζωή του, αν έχει χάσει τη ζωή του και οι περισσότεροι αυτό υποθέτουν, χρειάζεται να διεξαχθεί έρευνα. Πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να δούμε τι πραγματικά συνέβη και αν διεπράχθη ένα έγκλημα να βρούμε τους ενόχους. Θα πρέπει να βρούμε όλες τις πληροφορίες που μπορούμε. Η έρευνα υποστηρίζεται το ώστε να έχει επιτυχία. Δεν μπορεί να γίνει μία ανοιχτή, αλλά όλα θα γίνουν σωστά και αποτελεσματικά. Οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή για μας είναι σημαντική. Και αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του λαού, του κοινού. Πώς να διαχωρίσουμε πολιτική από επιχειρήσει. Αυτό είναι κάτι από το οποίο περιμένουμε άτομα από εσά από τους Ρουμάνους και από άλλους. Και θα είμαστε σοβαροί όσον αφορά την προσέγγιση μας. Δεν περιοριζόμαστε μόνο στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, δηλαδή πώς να απελευθερωθεί, να απορριθμιστεί η οικονομία, πώς να ακολουθηθούν οι αποτελεσματικότερες πρακτικές, δηλαδή να εισάγουμε τις καλές πρακτικές και στην ε, Ουκρανία. Ο, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως επισκέφθηκε τη Γεωργία πρόσφατα και είδε ότι έχουν πετύχει πολλά θετικά αποτελέσματα σχετικά με αυτό. Κάνουμε το ίδιο και εμείς παράλληλα, αλλά μαθαίνουμε από διάφορες πηγές πώς να απελευθερώσουμε την οικονομία. Η Ουκρανική κυβέρνηση έχει καταργήσει 90% των αδειών που έπιναν το αίμα των επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Όσον αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ, κινούμαστε προς ένα αυτόματο σύστημα επιστροφής του ΦΠΑ που θα εφαρμοστεί στο μέλλον και ξέρουμε ότι είναι ένα οξύ πρόβλημα αυτό. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εάν δεν απάντησα σε όλες τις τεθήσεις ερωτήσεις. Δεν θέλω να ε, εκμεταλλευτώ το χρόνο σας. Ξέρω ότι έχετε ένα πολύ σημαντικό ομιλητή που θα ακολουθήσει, που είναι πολύ σημαντικό για την Ουκρανία. Μπορεί να απαντήσει σε πολλές από τις δικές σας τις ερωτήσεις που θέσατε. Γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η κατάστασή μας, έχει τις δικές του απόψεις. Ο, κύριος Επίτροπος που δεν α, ταιριάζουν απόλυτα τις δικές μου απόψεις, αλλά καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες που υπάρχουν. Εκτιμούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν να έχουμε ανταλλαγή απόψεων μαζί σα, να είναι ελεύθερη και ανοιχτή συζήτηση μαζί σα, που πιστεύουμε ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει σαν τελικό αποτέλεσμα να έχει την ε, βελτίωση βελτίωση της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής ζωής στην Ουκρανία και να υπάρξει μεγαλύτερη αποδοχή της ανάγκης να συμπεριληφθεί η Ουκρανία στην οικογένεια των ευρωπαϊκών κρατών συμμεριζόμαστε τις αξίες, ε, τις προσδοκίες, χρειαζόμαστε χρόνο, πρέπει να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες, ούτως ώστε να προσαρμοστούμε στα επίπεδα των όσων περιμένετε εσείς. Για, από μια αξιόπιστη και σημαντική χώρα της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ήταν μια συνάντηση πράγματι ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω αν δόθηκαν όλες οι απαντήσεις. Θα συνεχιστεί όμως ο διάλογός μας και θα υπάρξει δυνατότητα να συμπληρωθούν οι πληροφορίες, να ανταλλαγούν και άλλες απόψεις. Θα υπάρξει δυνατότητα να συνεργαστούμε και τόπου Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε στο επανειδήν. Δύο λεπτά διακοπή για να ακούσουμε μετά τον Επίτροπο τον κύριο Φούλε. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε, χρειαζόμαστε όλο το χρόνο. Δεν μπορούμε τίποτα να σπαταλήσουμε. Άλλωστε έφτασε εγκαίρος και ο Επίτροπος. Ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον φίλο και σημαντικότατο συνεργάτη μας, τον Επίτροπο Φίλε, με τον οποίο θα εξετάσουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπως είναι η αξιολόγηση και η αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας, που είναι μια διαδικασία που ήδη έχει αρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους. Είναι ένα πολύ βαρισίμαντο καθήκον και θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον Επίτροπο Φίλε εκ μέρους της Επιτροπής ότι Εκτιμούμε ιδιαίτερο στην προθυμία του για την τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητε του. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σημερινή παρουσίαση. Ήδη θυμάμαι την ακρόασή του πριν αναλάβει τα καθεκαντά του και την ψηφοφορία που τον επιβεβαίωσε στην ανάληψη των καθηκόντων του. Ήταν από τότε πολύ πρόθυμος για τακτικέ επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχίζει να είναι πολύ πρόθυμος, ε, ε, εξαιρετικά ικανός και ανταποκρίνεται στις, στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως έλεγα αυτή η συνάντηση προβλέπει τη συζήτηση όσον αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής, ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας όσον αφορά το άλλο θέμα με το οποίο ασχολείται ο Επίτροπος στη διεύρυνση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε στις 9 ε, Νοεμβρίου. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν, αν και είναι συναφή τα θέματα, να επικεντρωθείτε επί του πρώτου. Την περασμένη εβδομάδα έστειλα στους συναδέλφους το ερωτηματολόγιο που εσείς κύριε Επίτροπε μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο ε, στείλατε στα κράτη-μέλη και στα κράτη της γειτονίας, όπου εκεί τίθενται όσον αφορά το, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτή την πολιτική και κατά πόσο πέτυχαν το σκοπό τους, πόσο αποτελεσματικά ήταν. Η σημερινή συζήτηση με βέβαιος για όλους μας θα είναι μια ευκαιρία για προβληματισμό, ανταλλαγή απόψεων. Και θα, βάσει και των σχολείων που θα πορέων από αυτό το ρευματολόγιο και θα ενδιαφερόμαθα να σας ακούσουμε, να μας πείτε σχετικά με τους προσανατολισμούς που, που διεφάνισαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχατε στα... σε συζητήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών χθες νομίζω πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, θα σας δώσω αμέσως το λόγο και θα σας ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Θα σας απασχολήσω 10-15 λεπτά γιατί θα ήθελα πραγματικά να σας δώσω μια πλήρη εικόνα του τι κρύβεται πριν πίσω από την διαδικασία μεταρρύθμισης και για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Και όπως πάντα στην Επιτροπή σας, πάντα ε, θέλω να ακούσω και τα δικά σας σχόλια. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, είναι χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας για την ανταλλαγή αυτήν απόψεων για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία. Η Σύνθηκε της Λισαβόνας δημιουργήσε τους όρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί ένας παγκόσμιος ε, παράγοντας. Διάφορες φορές ε, εδώ στο Κοινοβούλιο έχω δηλώσει ότι ως Επίτροπος για Διεύρυνση και την Γειτονία σκοπεύω να συνεργαστώ στενά με την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο και την Υπηρεσία εξωτερική δράση για να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εκπληρώσει αυτή τη φιλοδοξία τη. Να πω ωστόσο ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να καταστεί αξιόπιστος παγκόσμιος παράγοντας θα πρέπει να ξεκινήσει από την γειτονιά της, από την από χώρε. όμορες χώρες. Τους επόμενους ε, ε, μήνες και τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να καταδείξουμε την δυνατότητά μα να δράσουμε με πιστικό τρόπο σε ό,τι αφορά την πολιτική γειτονία και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και όλες τις ευκαιρίες που έχουμε που μας προσφέρονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας και θα αποτελέσει αυτό ένα από τα βασικά ορόσημα βάσει των οποίων θα κριθεί η εξωτερική μας πολιτική και η εξωτερική πολιτική και σχετικές διατάξεις της συνθήκης Λισαβόνας. Αυτό κάνει την ε, στρατηγική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ένα πολύ επίκαιρο εγχείρημα. Βρισκόμαστε το μέσο της διαδικασίας διαβούλευσης. Έχουμε λάβει α, τα σχόλια σχεδόν όλων των κρατών μελών και των χωρών που συμμετέχουν στην πολιτική γειτονία. Έχουμε ακούσει τους εμπειρογνώμονες, τους ακαδημαϊκούς. Έχουμε συναντηθεί με τους ανώτερους ε, αξιωματούχους των χωρών εταίρων αυτές, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη, τα κρατημέλη, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και σήμερα βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Σε δέκα ημέρες θα συνδυθώ με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλες τις ε, περιοχής. Δεν μπορούμε ακόμα να εξαγάγουμε συμπεράσματα, αλλά θα πρέπει να εντοπίσουμε κάποια θέματα τα οποία ανακύπτουν και τα οποία χρήζουν περαιτέρω ε, περισυλλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των εκθέσεών τους έχει στο παρελθόν συμβάλει σημαντικά για την ε, διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και είμαι σίγουρος ότι και σήμερα στη συζήτηση θα μας δώσετε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα εμπλουτίσουν τις περαιτέρω σκέψεις μας. Στην επιστολή που έστειλα την προηγούμενη, τον προηγούμενο Ιούλιο με την Κάθη Άστον προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ε, ε, Υπουργό Εξωτερικών των ε, χωρών εταίρων, έχουμε θέσει τρία ερωτήματα. Ποιο θα πρέπει να είναι το όραμά μας καταρχάς σε ό,τι αφορά την πολιτική γειτονία για τα επόμενα 10 έως 15 χρόνια. Ποιος, ποιοι θα πρέπει να είναι οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι που θα επιδιώξουμε ευρύτερα κατά τη διάρκεια της θητείας του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και κατά τρίτον πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα μέσα και τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Για να δοκιμάσω λοιπόν τώρα να απαντήσω στις ερωτήσεις αυτές, να ξεκινήσω από το όραμα. Να πω ευθύς εξ αρχής ότι όλοι μας οι εταίροι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ευρή αυτή διαδικασία διαβούλευσης. Όλοι θέλουν πιο στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει υψηλού πολιτικού διαλόγου. Όλοι οι εταίροι ανυπομονούν και θέλουν μεγαλύτερη οικονομική ενσωμάτωση βάσει της προσέγγισης της νομοθεσίας και της ε, σύγκληση των κανονισμών, προκειμένου να καταστεί πιο εύκολη η κινητικότητα και να αυξηθεί η οικονομική συνεργασία. Υπάρχει μια σαφής ε, έκκληση για μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική γυμνίασης. Ακόμα και αν πολλές χώρες, ε, πολλοί από τους εταίρους, ε, δεν προτιμούν, αν θέλετε, και δεν τους αρέσουν κάποιες επιμέρους διατάξεις. Είχατε μια τέτοια συζήτηση πριν από λίγο. Αυτό είναι φυσικά πολύ θετικό, αλλά δεν είναι αρκετό απαραίτητα. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε μοναδικοί παράγοντες στην πολιτική γειτονία και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι επιδιώκουν να επεκτείνουν τη σφαίρα επιρροή του και μάλιστα με έναν τρόπο το, ο οποίος δεν είναι πολύ συμβατό συμβατός με τις ευρωπαϊκές αρχές ή με το κεκτημένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λευκορωσία συμφώνησε να κάνει Τελωνιακή Ένωση με τη Ρωσία, ενώ η οικονομική και πολιτική επιρροή της Κίνας αυξάνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφής σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες της προς τους ε, γείτονε τη, γιατί θεωρώ ότι δεν ήμασταν πάντα τόσο σαφείς όσο θα έπρεπε. Η αντίδρασή μας, η απόκρισή μας, αν θέλετε, στις ε, απαιτήσει που τίθενται από τους ε, γειτονέ μα, ιδιαίτερα στην περιοχή τη Μεσοδίου, σε κάποιε περιπτώσει έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στου τύπου παρά στην ουσία. Θα πρέπει η προσέγγιση μα, μάλλον η προσέγγιση μα συχνά προ διάφορε χώρε δεν ήταν τόσο α, συνεκτική και ενιαία. Θα πρέπει να τονίζουμε πάντα τις κοινέ αξίες. Θα πρέπει με μεγαλύτερη έμφαση να τονίζουμε ότι η καλή διακυβέρνηση και η πολιτική μεταρρύθμιση δεν αποτελούν, αν θέλετε, προαιρετικά στοιχεία της πολιτικής μας, αλλά ότι συμβαδίζουν ε, ε, άρεκτα με τις ε, πιο έντονες πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω ενός δικτύου διμερών και πολυμερών επαφών με τα κοινοβούλια των χωρών εταίρων, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση των δημοκρατικών αρχών. Οι διαβουλεύσει μας ω τώρα έχουν καταδείξει ότι υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό ομοφωνία σε ό,τι αφορά το όραμα της πολιτικής ε, γειτονίας. σύμφωνα και με το άρθρο 8 της ε, Σύνθηκης της Λισαβόνας προκειμένου η πολιτική συνεργασία και η οικονομική συνεργασία να είναι όσο πιο βαθιά γίνεται. Πόσο στενή τώρα θα είναι αυτή η συνεργασία. Όπως είπε και ένας εμπειρογνώμονας, ο μακροπρόθεσμος στόχος θα μπορούσε να ανταποκρίνεται σε οτιδήποτε μεταξύ μιας σφαιρικής και σε βάθος ε, ε, περιοχής ε, ελευθέρου εμπορίου, συν 1% και μείον 1% ανάλογα φυσικά και με τους μεμονωμένους ε, εταίρους. Σε ό,τι αφορά την οικονομική ενσωμάτωση τώρα, την οικονομική ενοποίηση, αυτό μας ε, οδηγεί ουσιαστικά σε μια πλήρη ένταξη στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και στην επέκταση των τεσσάρων ελευθεριών που απαιτούνται για την υιοθέτηση του κοινωνικού κοινοτικού κεκτημένου. Και εδώ υπάρχουν κάποια σημαντικά χάσματα μεταξύ των ε, προσδοκιών των εταίρων και μεταξύ αυτών που προτίθεται να διαθέσει, να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο χάσμα έχει να κάνει με τον αριθμό των ελευθεριών, των οποίων απολαμβάνουν οι πολίτες των χωρών εταίρων, γιατί οι εταίροι μας ε, θεωρούν ότι θα πρέπει να έχουν και τις τέσσερις ελευθερίες, ενώ κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, περιορίζονται σε τρεις από τις τέσσερις βασικές ε, ελευθερίες και είναι σαφείς και ανησυχούν με καταμετρό τρόπο πρέπει να προσθέσω σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ε, κίνησης. Το δεύτερο έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση, γιατί οι εταίροι μας τονίζουν το κόστος των μεταρρυθμίσεων που προκύπτει από την σύγκληση με το κοινωνικό κεκτημένο και κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλουν, ε, διστάζουν να συζητήσουν τους ε, πόρους που χρειάζονται για την ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων. Ίσως να χρειάζεται μια βαθμιαία προσέγγιση και μια πιο σαφή, αν θέλετε, διαφοροποίηση, μια DCFTA, μια πιο σφαιρική δηλαδή και πιο σε βάθος ε, περιοχή ελευθέρου εμπορίου και ένα καθεστώς χωρίς ε, θεωρήσεις δεν αποτελούν μόνο σαφές δεσμεύσεις για τους ε, χώρες εταίρους, αλλά εκπροσωπούν και προϋποθέτουν μάλλον και ότι υπάρχει και η διοικητική δομή για να εκπληρωθούν αυτές οι ανάγκες. Θα πρέπει να ανταμείβουμε όμως την πρόοδο όπου σημειώνεται. και θα πρέπει οι χώρες αυτές οι οποίες ε, κάνουν πραγματικά πολιτικές μεταρρυθμίσεις ή εφαρμόζουν τέτοιες ζώνες ελεύθερου εμπορίου να ε, λαμβάνουν και τα απαραίτητα κονδύλια. Δεν γίνεται αρκετή διαφοροποίηση στην παρούσα φάση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο άμεση σε ό,τι αφορά την ε, ελευθερία κίνηση των χωρών εκείνων που κάνουν πραγματικά ό,τι χρειάζεται στα εξωτερικά του σύνορα να πω στο σημείο αυτό ότι θεωρώ ότι η διαφοροποίηση θα πρέπει να βασίζεται και στις φιλοδοξίες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην προθυμία που έχουν για να αποδέχονται τις κοινέ αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, στην απόδοση τους σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση και τις μεταρρυθμίσεις και όχι στην γεωγραφική τους θέση. Φυσικά κάποιες από τις γειτονικέ χώρες ε, είναι ευρωπαϊκές και θεωρούν ότι θα μπορούσαν στο μέλλον να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι φιλοδοξίες αυτές δεν αποτελούν λόγο για να προσφέρουμε λιγότερα σε άλλες χώρες ή για να έχουμε λιγότερες απαιτήσει έναντι των χωρών αυτών. Αν ε, οι ευρωπαϊκές ε, γειτονικές χώρες είναι πιο φιλόδοξες, θα πρέπει να θέσουμε και τον πύχη πιο ψηλά. σχεδόν όλοι οι εταίρες συμφωνούν και σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι θα πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία να παραμείνει η ενιαία ομπρέλα, αν θέλετε, για τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας. Υπάρχουν διάφοροι τομείς στους οποίους θα πρέπει να δώσουμε προσοχή μέσω πρόθεσμα. Και βλέπουμε ότι επτά θέματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Ένα είναι το αίτημα διαφόρων εταίρων για πιο πολύ πολιτική καθοδήγηση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με, μια πιο με ένα πιο βελτιωμένο συνεχή διάλογο επί της ουσίας σε πολιτικό επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι λογικό αυτό το αίτημα, θεμητό και μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε παρανοήσεις και δύσκολα θέματα σαν να πνεύμα εμπιστοσύνης και εταιρική σχέσης. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να εφαρμοστεί και στην πράξη η ιδέα αυτή, όχι μόνο μεταξύ Υπουργών Εξωτερικών, αλλά και σε άλλους τομείς στενή συνεργασία. Δεύτερο θέμα που μας απασχολεί είναι τα DCFTAs, που αποτελούν, αν θέλετε, και τον πυρήνα της προσφοράς μας προοπτική συμμετοχή στην εσωτερική αγορά αποτελεί ένα βασικό κινητήριο μοχλό για την επιτευξή αλλαγών. Θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις για τα DCFTA βράχη πρόθεσμα να γίνονται με τους πιο προηγμένους ε, από τους γειτονές μας και στην Ανατολή και προς τον Νότο. Τονίζουν οι εταίροι μας πόσο σημαντική είναι η πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα. Επίσης, να τονίσουμε από πλευρά μα ότι προκειμένου οι εταίροι μας να μπορούν να αντρέψουν τους καρπούς μιας τέτοιας συμφωνίας, θα πρέπει να γίνουν και σοβαρές μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η δικαιοσύνη του δικαστικού σώματος και να καταπολεμηθεί η ίδια φθορά. Τρίτο θέμα, τρίτο αίτημα είναι η πιο εύκολη κίνηση των ε, πολιτών. Παρά τις πολιτικές δυσκολίες, ε, ε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα αιτήματα των εταίρων μας και θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο το ευρύτερο πλαίσιο. Να μην έχουμε μια προσέγγιση άσπρου ή μαύρου. Ίσως θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια πιο ευρεία προσέγγιση στην κινητικότητα και στην μετανάστευση. Μια προσέγγιση διπλού ωφέλους και προς τις δύο πλευρές. Ή να εστιάσουμε σε ορισμένες κατηγορίες ατόμων, για παράδειγμα φοιτητές, ε, ε, επιχειρηματίες, ερευνητέ ή να γίνει μια έντονη διαφοροποίηση, στην οποία αναφέρθηκα και προηγουμένως. Τέταρτο θέμα, οι παρατεταμένες ε, συγκρούσεις και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξευρεθεί λύση προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό το ερώτημα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Η ανυκανότητα συμβολής στην επίλυση συγκρούσεων τονίζεται συχνά ως ένα από τα βασικά ε, μειονεκτήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, γειτονίας παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά ξεπερνά την πολιτική αυτή. Οι εταίροι μας μας έχουν ζητήσει να είμαστε πιο δραστηροί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο έντονα παρούσα και να δίνει πιο πολλούς πόρους για την ε, οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Υπάρχουν κάποιες σαφές προσδοκίες από πλευράς των εταίρων μας με το πλαίσιο και τις συνθήκες της ε, Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει και την ΚΕΠΑ και την ΕΠΑ με πιο ενιαίο τρόπο. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε περαιτέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Ένας πέμπτος τομέας, μια πέμπτη έκκληση έχει να κάνει με την εμβάθυνση τη της τομεακής συνεργασίας. Υπάρχει τέτοια α, επιθυμία μεγαλύτερη συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η εκπαίδευση, η βιομηχανική συνεργασία ή η μεταφορά τεχνολογίας. Αυτό είναι και προς το δικό μας συμφέρον και θα πρέπει με θετικό τρόπο να ανταποκριθούμε. Επίσης, οι εταίροι μας θέλουν να συμμετάσχουν πιο έντονα, να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα και να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Ένα έκτο θέμα έχει να κάνει με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Οι οργανώσεις ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών, CSOs, στις ε, χώρες εταίρους, είναι ο πιο πιστός μας σύμμαχος σε ό,τι αφορά την πρόθεση των αξιών μας. Είναι επίσης σημαντικό σύμμαχο σε ό,τι αφορά την σύγκληση προς τα ευρωπαϊκά στάνταρ σε τομείς όπως το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να συμμετάσχουν και να τους εμπλέξουμε πιο έντονα στην διαμόρφωση και στην παρακολούθηση της πολιτικής. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση με τις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτές και να ενισχύσουμε τις ικανότητές τους. Τέλος, υπάρχει και το θέμα των περιφερειακών ε, χαρακτηριστικών στην ε, περιοχή γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια μεμονωμένη και ειδική, αν θέλετε, προσέγγιση στις διάφορες περιοχές ε, θα πρέπει να αποτελέσει τη βασική μας προσέγγιση. Είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας θα πρέπει να προωθήσει και την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των εταίρων μας ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ε, Ανατολικής Ιταρικής Σχέσης και της Ένωσης για τη Μεσόγειο, που αποτελούν τις βασικές, αν και όχι τις μόνες, ε, περιφερειακές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Με την ε, εταιρική σχέση προς Ανατολάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει μια φιλόδοξη ατζέντα για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις έξι χώρες εταίρους προς Ανατολάς και σε διμερές επίπεδο, αλλά και συνολικά. Οι σχέσεις αυτές οι σημαντικές και αυτή η πολυμερή συνεργασία έχουν καταστεί πολύ έντονες. Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας θα μας δώσει την ευκαιρία να εξετάσουμε τα πρώτα επιτεύγματα και να προετοιμάσουμε με ε, επιτυχία την Σύνοδο στη Βουδαπέστη τον επόμενο Μάιο. Η Ένωση για τη Μεσόγειο επίσης κινείται και εξέλισσεται θετικά παρά τις ε, πολιτικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την ε, διαδικασία ερήνευσης στην Μέσα Ανατολή. Η γραμματεία που θα δημιουργηθεί είναι σχεδόν έτοιμη να δημιουργηθεί και πολλά έχουν ήδη γίνει που θα ενισχυθούν από την Ένωση για την Μεσόγειο. Θα πρέπει να εντοπίσουμε πρακτικούς τρόπους για να συμβάλλουμε στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας αυτής και θα πρέπει να βοηθήσουμε προκειμένου να επιτευχθούν οι ουσιώδεις στόχοι σε ό,τι αφορά την ε, περιοχή της Μεσογείου τα επόμενα χρόνια. Τέλος, να έρθω στο θέμα των πολιτικών μέσων, των οικονομικών μέσων και τέλος των πόρων. Τα σχέδια δράση στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας έχουν ε, αποδείξει την αξία τους ως ένα κεντρικό εργαλείο μέσω εφαρμογής πολιτικής. Τώρα που έχουμε περάσει πλέον στη δεύτερη γενιά θα πρέπει να είναι πιο εστιασμένα τα μέσα αυτά, να υπάρχει καλύτερη σχέση με την μεταρρυθμιστική ατζέντα των χωρών εταίρων και με τους χρηματικούς πόρους που διατίθενται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και Τερικής Σχέσης αποτέλεσε μια βαθμιαία αλλαγή στον τρόπο που δίνουμε την ενίσχυσή μας. Πολλοί ωστόσο υπογραμμίζουν ότι πολλά θα πρέπει ακόμα να γίνουν για να υπάρξει πιο έντονη σχέση μεταξύ των προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και της οικονομικής συνεργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη ευελιξία για την ανταπόκριση στις ε, ανάγκες που ανακύπτουν. Επίσης, οι χώρες εταιρείς οι χώρες εταιρείς πολλές φορές μας ζητούν να κοιτάξουμε πιο πολύ το θέμα της ε, βοήθειας, της ενίσχυσης στη φάση πριν από την ε, ένταξη. Υπάρχει μία αντιστάθμιση μεταξύ, αν θέλετε, μια σχέση μεταξύ αποδοτικότητας και ελέγχου πάντα σας απασχολούν θέματα δημοκρατικού ελέγχου σε ό,τι αφορά τις ε, δαπάνες, τις εξωτερικές. Πάντα υπάρχει ο δημοκρατικός έλεγχος στα πλαίσια του, της πολιτικής γειτονίας, ο οποίος πάντα λειτουργήσε σωστά. Να σκεφτούμε λοιπόν πρωτού α, αλλάξουμε τη διαδικασία αυτή. για να μην καταστεί πιο δύσκολη η παροχή βοήθειας ή πιο επίσημη χωρίς ε, λόγο. Να τονίσω το εξής, ότι η ενίσχυση στις ε, χώρες ε, τις γειτονικές είναι διαφορετική επί της ουσίας δηλαδή σε σχέση με την κλασική αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει γρήγορα να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που ανακύπτουν και θα πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο υποχρεώσεων Διστάζω πάντα να μιλώ για τους χρηματοοικονομικούς πόρους σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, μπορούμε να συντονίσουμε την ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με καλύτερο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα σχέδια δράσης μας ως σημεία αναφοράς. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να δώσουμε και στα μέσα αυτά τα επαρκή κονδύλια. Δεν μπορούμε να ζητάμε εκτενής αλλαγής και από την άλλη να, στε, να αρνούμαστε να απορρίπτουμε την ε, ενίσχυση που χρειάζεται. Θα πρέπει να θέσουμε ως προτεραιότητα στην επόμενη χρηματοοικονομική περίοδο την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Να κάνω κάποια καταλεκτικά σχόλια. Σας ε, ανέφερα κάποιες σκέψεις για κάποια θέματα τα οποία ανακύπτουν από την στρατηγική αναθεώρηση. Πρόκειται για κάποια προκαταρτικά σχόλια, τα οποία θεωρώ ότι θα εξελιχθούν στην πορεία, θα καταστούν πιο συγκεκριμένα όσο συνεχίζεται και τη δικασία διαβούλευσης. Την 1η Φεβρουαρίου η κυρία Άστον και εγώ θα καλέσουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τις χώρες εταίρους σε μια υπουργική σύνοδο και θέλουμε να προκύψει μια κατευθυντήρια γραμμή, μια καθοδήγηση για τις προτάσεις που θα υποβάλουμε τον Απρίλιο σε ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήθελα ωστόσο να σας αναφέρω κάποιες αρχικές σκέψεις σήμερα, να ακούσω και ποιες είναι οι δικές σας ε, αντιδράσεις και προτάσεις. Γιατί αν θέλουμε η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία να καταστεί μια άγκυρα για τους ε, γείτονές μας και έτσι να αντικατοπτρίσετε τις φιλοδοξίες της ε, συνθήκης, χρειαζόμαστε και τις δικές σας απόψεις και την δική σας ενίσχυση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ε, Επίτροπε Φιούλε. Ο κύριος Μπροκ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας πω το εξή. Εδώ και καιρό, μάλλον και πρώτη φορά εδώ και καιρό, έχω την εντύπωση ότι προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά με μια σαφή στρατηγική. Με μια σαφή στρατηγική που έχει και ένα επιχειρησιακό σκέλος. Γιατί ως σήμερα ξοδεύαμε πολλά χρήματα, τα οποία όμως δεν είχαν μια συγκεκριμένη στοχοθέτηση. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στο παρελθόν. Και θυμάμαι τον ε, προκάτοχό σας, μάλλον θυμόμενος τον προκάτοχό σας, ε, ενισχύεται αυτή η εντύπωση που έχω. Χαίρομαι που θα συνεργαστούμε στενά για να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Και πολλές φορές σε πολλές εκθέσεις πραγματευθήκαμε τέτοια ερωτήματα όπως αυτά που θέτετε κι εσείς. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική. Είναι εξίσου σημαντική η, ευρωπαϊκή, η ανατολική πτυχή και η ε, νότια πτυχή. Απλά η διαφορά είναι στην μέθοδο. Και αυτό έχει τις ανάλογες συνέπειες. Γι' αυτό λοιπόν είμαι περίεργο. για το... Είμαι... Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το προωθήσουμε. Και είχε πει η Ρωμάνα Πρόντι ότι υπάρχουν όλα εκτός από τους θεσμούς. Δηλαδή να δούμε τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις για την ε, ζώνη ελευθέρου εμπορίου, για την πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Πώς μπορούν να καταστούν κάποιες χώρες μέλη της, ε, του Σέγγεν χωρίς να έχουν γίνει μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά άλλα. Ο Ευρωπαϊκός ε, Οικονομικός Χώρος να καταστεί το υπόδειγμα. Αυτό δεν μπορούν να είναι ίδια σε ό,τι αφορά την μέθοδο, αλλά για να έχουμε μια γενικότερη ιδεολογική προσέγγιση να υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική για να μην ε, κλείσουμε την πόρτα στους εταίρους μας, αλλά ούτε να υπερφορτώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Παντσέρι για δύο λεπτά. Ο κύριος Παντσέρι, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κ. Μπρόκ. Συμφωνώ μαζί του και σε αυτά που είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ όσον αφορά τον Επίτροπο για το πόσο διαθέσιμο είναι και πόσο δείχνει θέληση που δεν είναι κάτι κοινό σε όλους του επιτρόπους και για αυτά που είπε προφανώ. Συμφωνώ και με αυτά. Έχω να θέσω κάποια σύντομα ερωτήματα. Η πολιτική γειτονία σαν αμφισβήτητα είναι κάτι στατηγικό. Χρειάζεται ένα γενικό όραμα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονία. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει σήμερα να προσανατολιστούμε ίσως με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να κάνουμε προσπάθειες και να δώσουμε και χρήματα προς τον Νότο και προς τη Μεσόγειο. Είναι προφανής σχεδόν οι, ε, λόγοι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που δημιουργούνται εκεί, αλλά και από εκεί προέρχονται και πολλές λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματά μας. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα. Χρησιμοποίησατε ισχυρού λόγους του συμμερίζομαι. Έχουμε πει πολλά, δεν έχουμε δώσει ουσία και να δώσουμε ουσία δεν σημαίνει μόνο χρήματα, αλλά πάνω απ' όλα σημαίνει να δώσουμε μεγαλύτερα, μεγαλύτερους όρους και δεσμούς εναντί αυτών των χωρών για τη δημοκρατική διαδικασία. Μιλήσατε για οικονομική ολοκλήρωση. Ε, πολλές χώρες ζητάνε μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα, περισσότερο από τους οικονομικούς πόρους, που είναι σημαντικοί προφανώς, οικονομικοί πόροι, διότι είναι χρήσιμοι για την επιτύχηση των στόχων, πάνω απ' όλα όμως ζητούν δημοκρατικές, υλικές και άειλες υποδομές. Όπως εκπαίδευση αυτή τη δημοκρατία, το θέμα της, στο θέμα της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να του ρίξουμε μια ματιά αυτού του θέματος και κατά την άποψή σας ίσως θα πρέπει ε, να επιλέγουμε καλύτερα τους στόχους της χρηματοδότησης. Όσον αφορά την ε, στρατηγική που ακολουθούμε, εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω την, ε, το ρόλο του κάθε επιτρόπου. Αλλά ο ρόλος σας σχετίζεται όλο και περισσότερο με ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι η μεταναστευτική πολιτική. Βλέπω ότι υπάρχει διέρεση μεταξύ τη Επιτροπή Ελευθεριών και τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Υπάρχει και εδώ, υπάρχει αυτή η διέρεση και πολύ συχνά συζητάμε θέματα πολύ... και υπάρχουν μεγάλε διαχωριστικέ γραμμέ και ίσω είναι καλύτερα αν υπάρχει λίγο πιο σφαιρική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Η κυρία Νέιτ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σα συγχαρώ και να σας επενέσω για την έναρξη αυτής της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Και σας ευχαριστώ επίσης για τον τρόπο με τον οποίο μας παρουσιάσατε τις θέσεις σας και τις αντιδράσεις των κρατών μελών ως προς το ερωτηματολόγιο που τους στείλατε καθώς και στους εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Ίσως από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δημιουργηθεί μια βάση για αυτή την πολλά αναμενόμενη και απαραίτητη αναθεώρηση. Γιατί υπήρξαν πολλές αμφισημίες και αοριστίες ως προς τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Πιστεύω επίσης ότι εξακολουθούν να ισχύουν πολλές παρεξηγήσεις ως προς το θέμα αυτό. Και μερικές φορές υπάρχουν και αντικρουόμενες ε, προσδοκίες. Για παράδειγμα, εγώ προβληματίζομαι που πολλές ε, χώρες της ε, πολιτικής γειτονίας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί πολλά αλλά προσφέρει λίγα. Και αυτό θα αυτή η τακτική θα πρέπει να σταματήσει αν ε, επιδιώκουμε πρόοδο. Επίσης ήθελα να σχολιάσω τρεις επιμέρους πτυχές της πολιτικής γειτονίας. Καταρχήν το θέμα της ε, ελεύθερης διακίνησης ή της κινητικότητας. Είναι προφανές ότι όσο πιο αυστηρή είναι η πολιτική μας για τις θεωρήσεις, όλο και περισσότερες είναι οι απόπειρες παραβίασης ή ε, αναζήτησης εναλλακτικών μεθόδων παραμερίζοντας το θέμα των θεωρήσεων. Μερικές φορές έχουμε το σύστημα αυτό που λέμε revolving θεωρήσεις, δηλαδή πολύ βραχές θεώρησεις και διαδοχικές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα των θεωρήσω. Βλέπω το ρολόι σας που μου δείχνετε επιδεικτικά κύριε Πρόεδρε, αλλά το ζήτημα το θεωρήσω είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα του ανοίγματο των αγορών. Εκεί όντως θα πρέπει να δεχθούμε περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από τις χώρες αυτές, εταίρους της πολιτικής γειτονία. Το τρίτο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με όλες τι τις ε, να κάνει ό,τι μπορεί για να επιληθούν αυτές οι παγωμένες συγκρούσεις. Κύριε Σούλτς, για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που σας ευχαρίστησαν για την ενημέρωση που μας κάνατε σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε όλα τα σημεία που αναφέρατε και θεωρώ ότι θα πρέπει να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες και μάλιστα προς την ανατολική κατεύθυνση. Αλλά στον τίτλο σας είσαστε υπεύθυνος και αρμόδιος και για θέματα διεύρυνσης. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε μια σαφή, ένα σαφή προσανατολισμό προς τις χώρες εταίρους μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή και τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η προοπτική να κάνουν κάποιες χώρες πολιτικές μεταρρυθμίσεις ε, για να ενταχθούν τελικά κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι πολύ παραπλανητική. Το δίκτυο, αν θέλετε, έντονων σχέσεων συνεργασίας αποτελεί μια πιο ε, ρεαλιστική λύση, μια ε, ζώνη ελεύθερου εμπορίου σε βάθος, η συμμετοχή στο Σέγγεν, στη ζώνη Σέγγεν. Αυτό είναι πιο ρεαλιστικό από ότι μια παρουσίαση ατέρμονης, αν θέλετε, δυνατότητας ένταξης. Θα πρέπει λοιπόν η συζήτηση αυτή για τα όρια απορρόφησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην παραταθεί περαιτέρω μετά από τις συνθήκες Λισαβόνας. Σας ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Μέιερ για δύο λεπτά. Κύριος Μέιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο. Θυμάμαι στην πρώτη σας παρουσία εδώ. Συζητήσαμε για τους μηχανισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και τη Συμφωνία Σύνδεσης και μιλήσαμε για την ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης του άρθρου 2, του άρθρου 2 επαναλαμβάνω, ώστε όλες οι συμφωνίες σύνδεσης ε, να εξαρτηθούν από την αυστηρή τήρηση και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων των διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είχαμε συμφωνήσει από ό,τι θυμάμαι τότε στην ανάγκη εμβάθυνσης αυτού του μέσου για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, γιατί το άρθρο 2 δυστυχώς μένει ανεφάρμοστο σε θέματα πολιτικής γειτονίας και στην Μεσογειακή Λεκάνη. Το κράτος του Ισραήλ, για παράδειγμα, δεν εφαρμόζει το άρθρο 2 στη Συμφωνία Σύνδεσης και θα θυμάστε ότι την περασμένη εβδομάδα στην επικράτη της Δυτικής Σαχάρας έλαβε χώρα μια δολοφονία ουσιαστικά ενός 14χρονου ανήλικου Σαχαραουίτη από το Μαροκινικό στρατό. Το παιδί αυτό που προσπαθούσε να φτάσει στον καταβλισμό των Σαχαρουιτών που εγκατέλειψε τις πόλεις τους και μένουν σε καταβλισμούς εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους κατά του βασιλείου του Μαρόκου εις βάρος του δικαιώματος αυτοδιάθεσης όπως αναγνωρίστηκε από το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν ο Μαροκινός στρατός ε, θέρισε μια ανθρώπινη ζωή ενώ ταυτόχρονα ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ εκφωνούσε ομιλία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοινώνοντα το δεύτερο ανεπίσημο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης του Μαρόκου και του μετόπου Πολυσάριο προκειμένου να διαθετηθεί η σύγκρουση. Βέβαια, το Μαρόκο δεν τήρει τις υποχρεώσεις του στα κατεχόμενα εδάφη, ενώ υπάρχει και κρεμία αλληλευτική συμφωνία με το Μαρόκο. Για το συγκεκριμένο αυτό σημείο, ενώ πρόσφατα έχουμε και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, νομίζω ότι είναι η στιγμή κατάλληλη να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το άρθρο 2. Θα μας χρησιμεύσει τίποτα αυτό το άρθρο 2 στη συμφωνία σύνδεση ή θα μείνει τελείως αναξιοποιητό. Ευχαριστώ κύριε Μέιρ. Του ΣΥΠ για δύο λεπτά. Ο κύριος του ΣΥΠ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την γενική αυτή επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα επτά σημεία που προσδοκούν οι εταίροι μας. Νομίζω είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε τις προσδοκίες των εταίρων μας, των παραληπτών αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και ιδιαίτερα της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Έχουμε και τις προσδοκίες που σχετίζονται με την βοήθεια που περιμένουν οι χώρες αυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διαθετήσουν αυτές τις παγωμένες όπως τις αποκαλούμε συγκρούσεις. Δυστυχώ δύσκολα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πρόοδο στην περίπτωση της Μολδαβίας, της Γεωργίας, του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δεν υπάρχουν απτά παραδείγματα ε, για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πρόοδο στις παγωμένες συγκρούσεις ε, χάρη στην πολιτική γειτονία. Θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση κύριε Επίτροπε, κατά τη δική σας εκτίμηση το θέμα της κινητικότητας ή η ευκολότερη πρόσβαση στις θεωρήσεις. Για ποια χώρα ισχύει από τις γειτονικέ μας, ποιες από τις χώρες της πολιτικής γειτονίας βρίσκονται πιο κοντά σε πρόοδο και μπορούν να περιμένουν ότι χάρη στις εργασίες τους, στις δραστηριότητές τους, στις ε, αλλαγές που έκαναν μπορούν να περιμένουν αυτή την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τη βελτίωση της κινητικότητας. Επίσης θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, οικονομικές επιβραβεύσεις για τις χώρες αυτές που είναι εταίροι της ανατολικής, ε, γειτονικής, ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Δεν ξέρω, δεν θέλω να αναφέρετε συγκεκριμένες χώρες, αλλά με ποια κριτήρια κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαμε να επιβραβεύσουμε οικονομικά ορισμένες χώρες ώστε να ενθαρρύνουμε και άλλους εταίρους να συμμετέχουν πιο δραστήρια σε αυτή την πολιτική. Eh, Σας ευχαριστώ και η Τζιπ Σεβερίν για δύο λεπτά. Ο κύριος Σεβερίν. Είναι... Είναι σειρά μου τώρα να συγχαρώ τον Επίτροπο για την πρωτοβουλία του, αλλά και για τα μέχρι τώρα επιτεύγματα και την υλοποίηση του οράματός του. Ήταν απαραίτητη αυτή η πρωτοβουλία, έγκαιρη, επίκαιρη και πολλά υποσχόμενη. Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία, δυστυχώς η συζήτηση αυτή δεν μας δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία να συμβάλλουμε ιδιαίτερα ούτε δίνει και σας την ευκαιρία να εκμεταλλεύετε τις δικής μας συστάσεις. Περιμένετε λοιπόν και την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάποιες συζητήσεις που θα γίνουν σε στενότερο κύκλο προκειμένου να εστιαστούμε σε συγκεκριμένα σημεία και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε κι εμείς στη γενικότερη συζήτηση σε επίπεδο αρχών πιστεύω ότι μια καλή σφαιρική πολιτική είναι το σημείο αφετηρίας για μια αγαστή πολιτική γειτονία. Πιστεύω όμως ταυτόχρονα ότι μια συνεπής πολιτική γειτονία προαπαιτεί μια συνεπή Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, η συνέπεια αυτή δεν θα πρέπει να είναι μόνο θεσμική, αλλά και διανοητική. Δεν μπορώ να να βρω καλύτερη λέξη, γιατί έχουμε διαφορετικές ευαισθησίες, ανομοιόμορφες παραδόσεις, γνώσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να δείξουμε μία ενιαία προσέγγιση της γειτονία. Δεν θα πρέπει μόνο η Ιταλία να ενδιαφέρονται για τη Μεσόγειο, οι νότιες χώρες να ενδιαφέρονται για τη Μεσόγειο, μόνο η Ρουμανία να ενδιαφέρεται για τη Μολδαβία ή η Πολωνία για την Ουκρανία, για παράδειγμα. Αυτό θα εξασφαλίσει και καλύτερη συνοχή στην προσέγγιση, αλλά θα χρειαζόμαστε φυσικά και μια πολιτική σταθερότητα. Ως θέμα αρχής, λοιπόν, χρειαζόμαστε μια σταθερή γειτονιά για να είμαστε και εμείς σταθερότητα και θέλουμε και μια ασφαλή γειτονιά για να είμαστε και εμείς πιο ασφαλείς. Φυσικά χρειαζόμαστε και δημοκρατικές γειτονικές χώρες για να υλοποιήσουμε την προηγούμενη παραπετούμενη ασφάλεια και σταθερότητα. Και τέλος κάτι που δεν αναφέρατε, την κοινή γειτονία. Ίσως αυτό περιπλέξει τα πράγματα, γιατί γειτον... μερικές γειτονικές χώρες δεν είναι μόνο δικοί μας γείτονες, είναι και γείτονες άλλων. Οπότε Πώ θα τι αντιμετωπίσουμε αυτέ τι χώρε ω αποκλειστικά Γειτονικέ χώρε οπότε θα έχουμε ανταγωνιστικότητα ή άμυλα με άλλους που επίση του έχουν γείτονε. Ή θα επιδιώξουμε κάποιε τριμερεί τριγωνικέ συνεργασίε ή διμερείς ορισμένες περιπτώσεις. Και πώ θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα και στον άλλο μεγάλο γείτονα των γειτονικών μας αυτών χωρών για να συνεργαστεί μαζί μας. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας στην χορήγηση του χρόνου. Ελπίζω πάντως ότι θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Σε ευχαριστώ και Σεβερίν. Γιούλαντ για δύο λεπτά. Κυρία Γιούλαντ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Φούλ, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Έχω ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα σχετικά με αυτά που είπατε όσον αφορά την έλλειψη προοπτικής, όσον αφορά την πολιτική γειτονία. Δηλαδή ότι κοιτάμε πολύ μακριά, κοιτάμε μόνο στις γειτονικές χώρες και συμφωνώ ότι αν δεν μπορέσουμε να τους δώσουμε μια σαφή προοπτική δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι αυτέ οι χώρε θα κινηθούν πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο βάθο όσον αφορά τι μεταρρυθμίσει. Όσον αφορά την εσωτερική πολιτική, θα ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσουν στου λαού του για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε αρκετά δαπανηρέ μεταρρυθμίσει ενώ δεν έχουν σαφή προοπτική. Υποστηρίζω λοιπόν την προθυμία σας να, υπάρχει, να υπάρχουν σαφέστες προπτικές. Συγκεκριμένο ερώτημα όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών. Είπατε ότι είμαστε πρόθυμοι να ανοίξουμε τις αγορές. Λέμε συνήθως μεγάλα λόγια προς τις γειτονικέ χώρες. Λέμε τα μεγάλα λόγια, αλλά όσον αφορά την πράξη, δεν γίνεται. Εγώ μιλάω για την ώρα για τη γεωργία. Βλέπουμε ότι στην πράξη δεν ξεκινάμε καν τις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο και θέτουμε νέα τεχνικής φύσεως που απαιτούμε από τη στιγμή που συμμορφωθούν με τα προηγούμενα. Του θέτουμε άλλους όρους μετά. Και στην περίπτωση της χώρας μου, μπορέσαμε να ξεκινήσουμε τουλάχιστον τις διαπραγματεύσεις και παράλληλα η χώρα συνέχιζε με την συμμόρφωση με τους όρους που είχαν τεθεί και με τις μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να στείλουμε εμείς ένα μήνυμα ότι πραγματικά θέλουμε να υπάρξει αυτή η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μετά αφού ολοκληρωθούν οι όλες οι διεργασίες. Ευχαριστώ. Μπράντερ για δύο λεπτά. Η κυρία Μπράτνερ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Φούλε. Λέει η κυρία Μπράτνερ. Πρώτα απ' όλα έχω να θέσω κάποια ερωτηματικά. Τι μπορούμε να προσφέρουμε όσον αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων, εκεί έχουμε εστιαστεί, αλλά ίσως είναι πολύ στενό αυτό το πεδίο, πρέπει να το διευρύνουμε. Θέλουμε να ανοίξουμε την αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσης, αυτά τα γερικά προϊόντα και τα κρουστιφαντουργικά και το χάλιβα. Πρέπει εκεί να συζητηθεί ειλικρινώς το ζήτημα. Και θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να συζητήσουν το θέμα με ειλικρίνεια. Και κάτι άλλο, το θέμα της παιδείας και πώς οι νέοι φοιτητέ, οι νέοι επιχειρηματίες θα μπορούν να έρχονται και να διαμένουν για ένα χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διευρύνουμε την προσφορά μας και να ξεφύγουμε λίγο από το στενό θέμα της, ε, των θεωρήσεων. Παρόλο που είναι σημαντικό, θα πρέπει να επαναξετάσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ζήτησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διάφορες ε, συμφωνίες που δεν εφαρμόζονται. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί γι' αυτό. Χρησιμοποιούνται ρήτε συμφωνίε, αλλά δεν εφαρμόζονται θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Μιλήσαμε για τις παγωμένες συγκρούσεις, όπως αποκαλούνται, είναι το δυσκολότερο πρόβλημα και κάτι άλλο για τη Λιβύη, για το πρόγραμμα για συνεργασία που υπογράψατε και εσείς και η Επίτροπος η κυρία Μάλστρομ. Διάβασα ότι ένα μέρος από τα 50 εκατομμύρια θα βγει από το μέσο για τη σταθερότητα. Αυτό δεν το βρίσκω σωστό. Θα ήθελα εξηγήσει. Από πού πραγματικά προέρχονται αυτά τα χρήματα και πώς μπορείτε να υπερασπιστείτε αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπράτνερ. Κούγκαν για δύο λεπτά. Ο κύριος Κούγκαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, όλοι σας επενούν. Και εγώ θα ακολουθήσω την ίδια γραμμή, αλλά θα ήθελα να πηχήσω και τα λόγια τα αρχικά του Προέδρου, που είπε ότι όλοι εκτιμούμε την ετοιμότητά σας να έρθετε. Δεν είναι μόνο ετοιμότης και προθυμία, έρχεστε και δίνετε πραγματικά τη δυνατότητα να σας μιλήσουμε. Παρακαλώ λοιπόν, μην το θεωρήσετε σαν πυρουέτα διπλωματική, αλλά εκτίμηση της προσέγγισής σας. Και ε, δεν κάνατε και λιγμούς και πυρουέτες απαντώντας στις ε, ερωτήσεις και στα σχόλια. Άλλη φορά ελπίζω να το αποδείξετε και αργότερα όταν θα αρχίσετε να δίνετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που σας θέτουμε τώρα. Εκτιμώ τις σκέψεις που μας παρουσιάσατε σήμερα διότι θεωρώ δεν ήταν απλώς οράματα που τα περιγράψατε. Δεν ήσασταν απλώς οραματιστής. Δεν αοριστολογούσατε. Το ερώτημά μου είναι μάλλον εύκολο και χαλαρό. Είστε σε επίτροπος για την ευρωπαϊκή πολιτική, για την διεύρυνση και για την πολιτική γειτονία. Πώς βλέπετε αυτές τις δύο πτυχέ του χαρτοφυλακίου σα, Είναι συμβατά τα δύο χαρτοφυλάκια. Αποτελούν ένα κομμάτι τη ίδια εικόνας, δύο κομμάτια της ίδιας εικόνας ή διαφορετικά κομμάτια που είναι δύσκολο να συγχωνευτούν. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η προσωπική σα άποψη πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Ο κ. Παλέτσκης για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θερμά ευχαριστώ για τις αφέστατες και πολύ περιεκτικές σας παρατηρήσεις. Πολύ διεξοδικές και τα σχόλια που ακούσαμε έδειξαν ότι πολλοί συνάδελφοι συμμερίζονται το όραμά σας και θα το, θα το υποστηρίξουν τουλάχιστον στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και χαίρομαι γιατί υπάρχουν πολύ θετικές προοπτικές ε, για την υλοποίηση όλων αυτών των προσανατολισμών. Έχω μια συγκεκριμένη και πανεύκολη ερώτηση. Πώς εκτιμάτε την ε, κατάσταση στη Λευκορωσία εν ώψη των εκλογών ε, της 19 Δεκεμβρίου αλλά και μετά. Η Λιθουανία με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία έχουν ετοιμάσει κοινέ προτάσεις ε, για την ανατολική εταιρική σχέση προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία σε θέματα ενέργειας, μεταφορών και πολιτισμού. Πώς εκτιμά τα σχέδια αυτά και τις κοινέ προτάσεις των τριών χωρών, πώς θα μπορούσε να τις υποστηρίξει ηθικά, αλλά όχι μόνο ε, ηθικά, και πώς ε, αξιολογείται την πρόσφατη επίσκεψη της Λιθουανής Προέδρου Θάλια Γκριμπαουσκάιτε στο Μίνσκ. Σας ευχαριστούμε, κύριος Πέτερλε, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά που συναντιόμαστε αυτή την εβδομάδα και σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε συνεδρίαση και μας κάνατε την παρουσίασή σας. Μιλήσατε για τη φιλοσοφία αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χαρακτηρίσατε ως ε, σκεπή. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα ήθελα να επιμένω σε ορισμένα ζητήματα. Νεολαία, πρώτο θέμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κάποια κοινά προγράμματα ανταλλαγή νέων, ε, φοιτητών, ερευνητών κτλ. Δεύτερο ζήτημα, η κινητικότητα. Θέλουμε περισσότερη οικονομική συνεργασία, περισσότερη ανταλλαγή ε, γνώσης, μεγαλύτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Τουρκία, για παράδειγμα. Ασχολήθηκα με το θέμα αυτό την περασμένη εβδομάδα. Οι Τούρκοι επιχειρηματίες περιμένουν εβδομάδες ολόκληρες για να αποκτήσουν θεώρηση. Η κατάσταση αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Επίσης, θέμα υγείας και υγειονομικής κατάστασης. Και εκεί μπορούμε να ενισχύσουμε την συνεργασία γιατί υπάρχουν κάποιες ε, κοινέ ε, φιλοδοξίες για θέματα υγείας, όπως είναι η καταπολέμηση ασθενειών σαν τον καρκίνο ή κάποιες ανταλλαγές σε θέματα ε, αναπτυξιακά. Σε όλα αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαμε να έχουμε εκείνη προσέγγιση με τους εταίρους, γι' αυτό και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη κινητικότητα και στα θέματα της γνώσης, γιατί η γνώση δεν είναι μονόδρομος, αλλά διπλής κατεύθυνσης δρόμος. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πέτερλε, κυρία Γκόμες έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Επίτροπε. Δεν είναι μόνο οι γείτονε αυτοί που θέλουμε να επηρεάσουμε εκείνους που δεν έχουν τις ίδιες αξίες με μας. Καμιά φορά λησμονούμε και εμείς οι ίδιοι τις αξίες μας όπως είναι η έλλειψη στρατηγική όσον αφορά τι θεωρήσει και οι συμφωνίε επανεισδοχή με δικτατορίε που προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε μαζί τους. Και σχετικά με αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι δική σας ευθύνη, αλλά λυπούμεθα διότι μέχρι τώρα δεν βλέ, είδαμε ποιοι είναι οι όροι της συμφωνίας πλαισίου που διαπραγματευτήκατε με τη Λιβύη παρόλο που φεύγει την επόμενη εβδομάδα την προσωπία για τη Λιβύη. Καλωσορίζω την στρατηγική σας σκέψη και προσέγγιση και το ερωτηματολόγιο. Αλλά οι υπουργοί μας είναι πολύ καλά όσον αφορά τη στρατηγική ρητορική. Το θέμα είναι άμα αυτή η στρατηγική πρέπει να υλοποιηθεί σε δράση. Άρα θα ήταν χρήσιμο όταν τίθενται ερωτήματα. Ποια είναι η θέση τους επικρισίμων ζητημάτων, όπως είναι η σύγκρουση στην Κύπρο, που υπονομεύει όχι μόνο τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, αλλά και την σχέση μας και την ΚΕΠΑ και Δυτική Σαχάρα, όπου και συμφέροντα δικά μας ασφαλείας διακυβεύονται διότι στην περιοχή της Σαχάρας αυξάνεται η τρομοκρατία και η σύγκρουση Ισραηλινών Παλαιστινίων και άλλα θέματα. Είναι πολλά ε, ζητήματα. Θα έπρεπε να ζητήσετε του υπουργού εξωτερικού να επικεντρωθούν επ' αυτών και όχι να μα δίνουν αυτέ τι ε, δικαιολογίε φτωχέ μα δίνουν για να μην αλαμβάνει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μα λένε είναι στα χέρια του ΟΗΕ αυτό το θέμα και νύπτουμε τα σχήρα μα ή εθελοτυφλούμε. Αυτά. Συγγνώμη, δεν μπορώ να παραμείνω για να ακούσω την απάντησή σας, αλλά θα μου διαβιβάσουν την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Κρέσλερ Ντόφλερ. Για δύο λεπτά κύριος Ντόφλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε να κάνω κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με αυτά που είπε και ο κ. Σούλτς, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει σε κάποια φάση να συζητήσουμε και τα όρια της απορρόφησης. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θυμάμαι ότι ο Γιος Φίσερ είχε πει κάτι σχετικό πριν από κάποια χρόνια. Αν υπάρχει μια τέτοια, κάποια τέτοια όρια, αυτό τι σημαίνει, ότι κλείνουμε τη διαδικασία αυτή για πάντα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σήμερα, σε, δεν ξέρουμε σήμερα τι θα γίνει σε 30 χρόνια από τώρα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να το πραγματευτούμε το ερώτημα αυτό και προς το συμφέρον των πολιτών μας, οι οποίοι πλήττονται ουσιαστικά από κάθε ε, διεύρυνση. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και υπάρχει και ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Η εμβάθυνση είναι δυνατή μόνο ε, αν υπάρχει διεύρυνση. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλη και σίγουρη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο πιο πολύ μπορεί να προχωρήσει και η εμβάθυνση. Μπορούμε και αυτό να το συζητήσουμε και θα πρέπει να το συζητήσουμε να μην ασχοληθούμε μόνο με το, άμεσο ερώτημα του πώς θα διαμορφωθεί το επόμενο κύμα διεύρυνσης, αλλά να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση των τελικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορεί να κάνει η Ένωση και τι θέλουμε να κάνει η Ένωση. Θα πρέπει να το θέσουμε το ερώτημα αυτό. Το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και κατά τη διάρκεια της ε, συνθήκης η οποία τελικά κατέληξε να είναι η συνθήκη της Λισαβόνας. Πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η συζήτηση. Είσαστε διατεθειμένος να την προωθήσετε προκειμένου να το θέσουμε, αν θέλετε, ως προτεραιότητα και της εξωτερικής διάστασης, αλλά και της ιστορικής διάστασης. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Συγγνώμη, ο Επίτροπος, ο κ. Φούλα, έχει το λόγο για να δώσει μια απάντηση σε πολλές ερωτήσεις που σας ετέθησαν. Yeah, yeah. Uh, uh, I can make a choice, yeah. ε, μπορώ να κάνω μία επιλογή. Θα αρχίσω εκεί που σταματήσατε εσείς. Εναπόκειται σε εσά βέβαια, αλλά εγώ είμαι υπέρ. Θα έχουμε το πακέτο της διεύρυνσης που θα λάβετε σε λίγες μέρες. Σήμερα δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε, αλλά σίγουρα θα ήθελα να γίνει συζήτηση όχι μόνο για τους όρους, για τις πολιτικές αιρέσεις της διεύρυνσης για το τι είναι εφικτό για την αντίληψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά να εξετάσουμε το κατά πόσο η διεύρυνση εξακολουθεί να είναι μια διαδικασία ενοποίηση της Ευρώπης ή έχει γίνει κάτι διαφορετικό και να δούμε τι σημασία έχει η διεύρυνση ως ε, μέσο που θα μας διευκολύνει στις πολιτικές μας. Ή να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύρυνση ε, για μια εποχή που πια το μέγεθος είναι σημαντικό αρχίζει και ξαναγίνεται σημαντικό. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα συζητήσουμε στα πλαίσια του πακέτου για τη διεύρυνση. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο και χρήσιμο. Και είναι σημαντικό το πλεονέκτημα που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια τέτοια συζήτηση. Γιατί δεν είμαι πάντα σε θέση να συζητώ αυτά τα θέματα με τους Υπουργούς Εξωτερικών, για παράδειγμα. για τη συμφωνία πλαίσιο. Η κάθε Άστον γνωρίζει το ζήτημα αυτό και γνωρίζει και τις συνέπειες της συμφωνίας πλαισίου που υπογράψαμε με το Συμβούλιο. Και πολλά κράτη στο Συμβούλιο εξέφρασαν επιφυλάξεις. Η κυρία Άστον εξετάζει αυτό το θέμα για να δει πώς μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εφαρμόσουμε τη δέσμευση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας πλαίσιο. Για τη Λευκορωσία. Δεν βλέπω μεγάλη πρόοδο εκεί. Περιμένουμε τις εκλογές. Οι εκλογές είναι ανέκαθεν μια ευκαιρία, είναι πάντα μια ευκαιρία. Τώρα θα είναι χαμένη ευκαιρία μετά τις εκλογές ή αν θα είναι ουσιαστική ευκαιρία, αυτό θα εξαρτηθεί από τις λευκορωσικές αρχές και φυσικά τους πολίτες της Λευκορωσίας. Εγώ σε καμιά δυο μέρες θα μεταβώ στο Μίνσκ για δεύτερη φορά και αυτή τη φορά κυρίως αποκλειστικά, καταρχήν δεν έχω συνάντηση με τον πρόεδρο στο πρόγραμμα, γιατί δεν είναι δόκιμο για έναν επίτροπο να, να συναντά πρόεδρο λίγο πριν τις εκλογές. Πάντως η Εθνική Πλατφόρμα είναι αυτή που στέλνει τον εκπρόσωπό της ε, στο δεύτερο φόρουμ ε, της κοινωνίας των πολιτών και εκεί θα επικεντρώσω τη συζήτηση στη Λευκορωσία. Ο πρόεδρος ε, Λουκασένκο γνωρίζει τις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι αξιώνει προκειμένου να προωθηθούν οι σχέσεις με τη Λευκορωσία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη θα εξετάσουν την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κοινό σχέδιο και δόθηκε το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο εντολής για τη διαπραγμάτευση της ε, Συμφωνίας Επανιστοχής και της Συμφωνίας ε, ε, διευκόλυσης των Θεωρήσεων. Κάτι που θα βοηθήσει τους πολίτες Λευκορωσίας να φτάσουν πιο κοντά σε αυτή την κινητικότητα της γνώσης. Μου άρεσε πολύ, κύριε Πέτερλε, η έκφραση που χρησιμοποίησατε. Επίσης, το θέμα δεν είναι να διαμορφωθεί οι συνθήκες για να προχωρήσουμε στις διμερείς σχέσεις, αλλά να έχουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε κατά πόσο υπήρξε μετρήσιμη πρόοδος από τις τελευταίες εκλογές και μετά. Και ελπίζω ότι θα υπάρξει πρόοδος και θα τηρηθούν οι δεσμεύσει που είχαν αναλυθεί από την τελευταία φορά που είχαμε εξετάσει το θέμα στη Λευκορωσία. Τώρα, από οικονομική άποψη, αργά ή γρήγορα η χώρα αυτή θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν πάντως αρκετές δυνατότητες συνεργασίες και το πλέγμα των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Λευκορωσίας είναι μια ιστορία χαμένων ευκαιριών ουσιαστικά μέχρι στιγμή. Σε αυτή τη στιγμή το μπαλάκι βρίσκεται στη Λευκορωσία, στο γήπεδο τη Λευκορωσίας. Εμεί είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα για να μπορέσει να αποκρούσει την μπάλα, να τη χρησιμοποιήσει, να την αποκρούσει και αυτό θα εξαρτηθεί από την προθυμία των ε, λευκορωσικών αρχών σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση και την πολιτική γειτονίας. Δεν είναι εύκολο να ασχολείται κανείς με 24 χώρες. Καθόλου εύκολο. Τώρα το... Αν μερικές φορές έχω πρόβλημα ως προς το διαχωρισμό αυτών των δύο κατηγοριών, δεν έχω ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Το είχα πει και στις ακροάσεις μου. Και δεν έχω αλλάξει γνώμη. υπάρχει μια σαφής ε, θεσμική διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ομάδων. Το είπα και προηγουμένως στην ε, ομιλία μου ότι υπάρχει και μια συμπληρωματικότητα σε ό,τι φορά τους μηχανισμούς, ε, τα μέσα αλλά και τους στόχους. Και εξαρτάται από εμά να αξιοποιήσουμε αυτά τα μέσα όσο καλύτερα γίνεται. Πάντως, δεν θα ήθελα πίσω από την πλάτη μερικών να γίνει η μεταφορά μιας χώρας από τη μία ομάδα στην άλλη. Αλλά όντως μερικές φορές είναι μια διανοητική πρόκληση. Συμφωνώ ότι για το μυαλό είναι σημαντική άσκηση γιατί είναι δύο διαφορετικές αυτές οι ομάδες των χωρών. Τώρα, συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω σταθερότητας. Και τέθηκε μία ερώτηση σε ό,τι αφορά τα κονδύλια για, την, για το αναπτυξιακό πρόγραμμα και τη συμφωνία με τη Λιβύη. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 50 συν 10 όχι συγγνώμη λέω επίτροπος, 40 συν 10. Αλλά δεν θέλω να σας παραπλανήσω, θα ενημερωθώ και θα σας απαντήσω γραπτός για το θέμα αυτό. Κοινοί γείτονε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω. Κύριε Σέβεριν, έφυγε στο μεταξύ ο κύριο Σεβερίν. Δεν είναι η πρώτη φορά που το αναφέρουμε. Το έχει ξαναθέσει αυτό το ζήτημα ο κύριος Σέβεριν. Πάντως, ευελπιστώ ότι για το θέμα αυτό θα λάβω κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές και προσανατολισμούς από την αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας. Και με το ενδιαφέρον δεδομένο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συζητήσουμε αυτό το θέμα και στην Επιτροπή. Από θεσμική και οικονομική άποψη υπάρχει μια σαφής γραμμή για το ποιες χώρες είναι εντός και ποιες εκτός πολιτικής γειτονίας, αλλά ταυτόχρονα οι χώρες αυτές δεν βρίσκονται εν κενό, βρίσκονται σε μια γεωγραφική περιοχή και επηρεάζονται από την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται και έχουν ενδιαφέρον για την περιοχή αυτή. Και φυσικά υπάρχει και αλληλεπίδραση με τις άλλες γειτονικέ χώρες και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Βέβαια το ζήτημα είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τους καλύτερους μηχανισμούς και τα μέσα στη διάθεσή της για να το κάνει. Πάντως ελπίζω ότι και με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Καθρινάστον θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα και με τους νέους μηχανισμούς της Λισαβόνας θα μπορέσει πιο αποτελεσματικά να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Κύριε Ξύπ, ε, θέλετε μια Ευρώπη που θα είναι πολύ πιο κοντά σε, ένα, σε μια απελευθέρωση των θεωρήσεων και εν καιρό σε μια απαλλαγή από κατάργηση των θεωρήσεων. Θα ακούσατε ε, και για το θέμα της διάσκεψης κορυφής με την Ουκρανία, θα σας το είπε ο για τις ε, Ουκρανίες, γιατί υπάρχει αυτή η πρόταση, κοινή πρόταση, για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να περάσουν στην επιχειρησιακή φάση του διαλόγου για τις θεωρήσεις και στην περίπτωση της Μολδαβίας. Καλό σημάδι αυτό και η Σεσίλια Μάνστρομ είναι πλέον αρμόδια επίτροπος για αυτό το θέμα, για αυτό το, σχέδιο, το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και φαίνεται σαν οδικός χάρτης. Παρόλο που το στοιχείο αυτό του μη αυτόματο χαρακτήρα ενισχύεται. Πάντως είναι ένας καλός οδικός χάρτης που μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε με σαφέστατο τρόπο ώστε να θαρρύνουμε συγκεκριμένες δράσεις και από τους εταίρους μας. Τώρα, ποια χώρα θα λάβει τους περισσότερους πόρους και την οικονομική επιβράβευση, αυτό το σημείο το κρατώ για την συνέχεια της συζήτησης, γιατί δεν έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Δεν θέλω να προεξοφλήσω κάποια, κάποια αποτελέσματα ευνοώντας ορισμένες χώρες. Πάντως, βλέπετε και στην Ανατολική Εταιρική Σχέση μια σαφή διαφοροποίηση για το πού πηγαίνουν τα κοινοτικά κονδύλια. Βλέπετε ότι κατά κεφαλή, να εξετάσετε το θέμα, η Μολδαβία είναι από τις πρώτες χώρες, ενώ η Λευκορωσία βρίσκεται ουραγός. Υπάρχει τεράστια διαφορά σε ό,τι αφορά τους πόρους. Δεν βλέπω άλλες συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί τα περισσότερα σχόλια αφορούσαν συστάσεις, ιδέες, προτάσεις, παρατηρήσεις, αλλά όχι ερωτήσεις. Και πραγματικά χαίρομαι, χαίρομαι που δεν έγινε απλώς ένας γύρος ερωταπαντήσεων ή μια ομοβροντία ερωτήσεων, ότι υπήρξαν και πολύ ενδιαφέροντα σχόλια και μαζί με τους συναδέλφους θα τα συμπεριλάβω στην διαδικασία αναθεώρησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το πιο σημαντικό σας σχόλιο ήταν οι τελευταίες παρατήσεις που κάναμε. Σας δείξαμε πόσο εκτιμούμε τη δέσμευσή σας, την αφοσίωσή σας στη δουλειά, πόσο θέλετε να συζητήσετε αυτά τα τόσο ευαίσθητα και σημαντικά θέματα μαζί μας. Μαζί με εσά θα τα καταφέρουμε και θέλουμε και εμεί να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Σα ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την παρουσία σα εδώ για την, τον επαγγελματισμό με τον οποίο συνεργαστήκατε μαζί μα και συνεργαζόσαστε και ελπίζουμε να συνεχιστεί ο διάλογος. Πέρα στη συνεδριά σα, θα ξαναρχίσουμε αύριο υπό την προεδρία του συναδέλφου Προβέρα στι 9 η ώρα το πρωί. Καλό σα βράδυ.